Καλημέρα σας, λέει ο Πρόεδρος. Καλώς ορίσατε εις την συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ξεκινούμε ευθύ αμέσως με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Πρώτα-πρώτα, θα σας πω ότι η ε, απογευματινή μας συνεδρίαση αναβλήθηκε για τις 7 Νοεμβρίου. Αν δεν έχετε κάποια ένσταση, έχω τώρα κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα πρώτα όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς των εργασιών μας. Έχουμε διερμηνία για κάποιες γλώσσες, όχι για όλες, τα έχουμε δανέζικα, φιλανδικά, μαλτέζικα, κροατικά. Ευχαριστώ την κατανόησή σας. Αυτό λόγω των περισμών από το, τη ταξία της αίθουσας. Επίσης, πρέπει να εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών, που είναι οι εξή. Πρώτα-πρώτα, ερωτήσεις προς Συμβούλιο και Επιτροπή, η εφαρμογή των, των ε, στρατηγικών και αποφάσισαν οι συντονιστές να υποβάλουν δύο ερωτήσεις προς Συμβούλιο και Επιτροπή από την ΛΥΜΠΕ και έχουμε κάποιες προφορικές ερωτήσεις που ήδη σας έχουν διανεμηθεί. Δεύτερον, έχουν προφορικές επιτροπές και επίσης ένα προφορικό ε, ψήφισμα για το πρόγραμμα δράσης 2014 για το e-justice, ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Και ε, εγκρίθηκε μια κοινή ερώτηση από τους συντονιστές ε, κοινή με την Επιτροπή Δικαιοσύνη Θα υποβληθεί στις 11 ε, Οκτωβρίου που θα γίνει η δεύτερη ολομέλεια, δεν έχετε κάποια ένσταση, αυτό εγκρίνεται και επίσης έγκριση των πρακτικών, αν δεν έχετε ούτε εκεί καμία ένσταση, πάμε παρακάτω στο σημείο 4. Η τρέχουσα κατάσταση των ενεξελίξεων διοργανικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Πρώτα-πρώτα, το τρίτο κοινό διάλογο για... Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και ακούγεται με ηχό ο πρόεδρος. Υπάρχει κάποια ε, παρεμβολή από το τηλέφωνο του πρόεδρου. Τώρα με ακούτε, λέει ο πρόεδρος. Ωραία, καλώς. Σήμερα έχουμε τον τρίτο κοινό διάλογο ε, για τις διαπραγματεύσεις τις οργανικές. Θεωρώ ότι θα κάνουμε βήματα λοιπόν πρόοδο σήμερα το απόγευμα όσον αφορά τις κατεξιοδότηση πράξης. Και άρα θα απεμπλακεί η υπόθεση και μετά τον τριμερή διάλογο θα ενημερώσω τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλς, για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις διαμετές αυτές για τα ζητήματα δικαιοσύνης. Η κυρία Μακοβέ είναι η εισηγήτρια και θα μας παρουσιάσει το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την οδηγία για τις κατασχέσεις. Κυρία Μακοβέη, έχετε το λόγο. Thank you, President. Uh, Μακοβέη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Από τότε που ψηφίσαμε και λάβαμε αυτή την ισχυρή διαμετρητική εντολή, συνεργαστήκαμε με την Λιθουανική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν τέσσερις πολιτικοί, τριμερείς διάλογοι, τεχνικές συναντήσεις. Προγραμματίσαμε και ένα άλλο τριμερή διάλογο για αυτό το μήνα, οπότε τα προβλήματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν αφορούν τα πιο σημαντικά ζητήματα όπως είναι η εκτεταμένη, η διευρυμένη κατάσχεση που δεν αφορά μόνο ποινικές υποθέσεις αλλά αφορά και κάποιες ειδικέ ε, περιπτώσεις αλλά και η κατάσχεση ισχυρα τρίτου. Έχουν γίνει μακρέ συζητήσει και επαφέ για τα σχετικά τριάρθρα με Συμβούλιο και Κομισιόν. Κατά τα λοιπά έχουμε συμφωνήσει. Ελπίζουμε ότι θα κλείσει η υπόθεση αυτή και θα έχουμε έναν αξιοπρεπή σύμβασμο πριν το τέλος του έτους και της Λιθωνικής Προεδρίας. Να ευχαριστήσω την κυρία Μπροσελίνα και την κυρία Αλφάνο για την συνεργασία τους και τους άλλους και οδησηγητές. Και να δούμε τι θα γίνει με το Συμβούλιο όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία σας προανέφερα. Θέλει κάποιο το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, ή το Συμβούλιο, η Επιτροπή για τις κατασχέσεις, το θέμα της κυρίας Μακοβέ, όχι, επομένως προχωρούμε στο σημείο υπαριθμών 5, που είναι η ενημέρωση στην Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή για την ενδεχόμενη αλλαγή έδρας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας της ΣΥΠΟΛ. και την περαιτέρω νομοθετική διαδικασία. Έχουμε κοντά μας, μάλλον βρισκόμαστε σε κατάσταση κατά την οποία η υπηρεσία αυτή η οποία πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο να καταρτίζει τους αστυνομικούς τώρα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η, το, η κυβέρνηση της χώρας είπε ότι το 2014 θα κλείσουν εκεί κατάσταση στον Μπράμφιλ και δεν προσέφεραν μια λύση. Το Μάρτιο η Επιτροπή πρότεινε να συγχωνευτεί η ΣΥΠΟΛ με την Europol. Συστήθηκε αυτή η πρόταση, υπήρξαν επιχειρήματα υπέρ και κατά. Έγινε συζήτηση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, οπότε τελικά το άτυπο Συμβούλιο του Ιουνίου στη Λιθουανία βεβαίως λόγω της Προεδρίας κάλεσε τα διευρώμενα κρατημέλη να υποβαλούν αιτήσει όσον αφορά την φιλοξένηση της ε, Αστυνομικής Ακαδημίας. Επτά κρατημέλη είπαν ότι ενδιαφέρονται, η Φιλανδία το Τάμπερε, η Ελλάδα για τη Βέρεια, η Ουγγαρία η πρόσφατη τη Βουδαπέστη, ε, η Ιταλία, τη Ρώμη, η Ιρλανδία, οι κάτω χώρες, τη Χάγη, την Άβυλα, η Ισπανία και στις 8 Δεκάτου το Συμβούλιο υιοθέτησε μια πρώτη τοποθέτηση όσον αφορά την Βουδαπέστη που θα είναι η προσωρινή έδρα της ΣΥΠΟΛ. Όμως, επειδή εδώ η διαδικασία που διέπει την κατάσταση είναι η συναπόφαση και έχουμε το άρθρο 4 της απόφασης του Συμβουλίου του 2005 η αλλαγή έδρας απαιτεί τροποποίηση της νομοθετικής πράξης όπως προβλέπει η συνήθεια της Λισαβόνας. Συναπόφαση. Άρα το Κοινοβούλιο εδώ έχει λόγο. Έχει. <clears throat> Λέγει δηλαδή το Συμβούλιο μόνο του δεν μπορεί να αποφασίσει. Άρα εξαρτάται και από εμά. κατόπιν συζητήσεως να κρίνουμε. ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να πούν κάτι όσον αφορά αυτή τη ε, διαδικασία. Όμως, πρώτα-πρώτα θα να τη γνώμη της Λιθουανικής Προεδρίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, και λυπή. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω για το θέμα αυτό, το οποίο σας παρουσίασε συνοπτικά ο Πρόεδρος. Και δεν θα πρέπει εδώ να επαναλάβω τα όσα ήδη ακούσατε. λόγω των περιστάσεων υποχρεωθήκαμε να αναζητήσουμε μια νέα λύση. Να τονίσω το εξή. Η κατάσταση προκλήθηκε από τη μονομερή απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να κλείσει τις εγκαταστάσεις του Μπράμσχιλ και επομένως η Προεδρία έπρεπε να διασφαλίσει ότι η Αστυνομική Ακαδημία η οποία είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της αστυνομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα πρέπει να μπορέσει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και έτσι αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, uh, η Λιθουανία ω τρέχουσα προεδρεύουσα ανακοίνωσε ότι μπορεί να δεχτεί υποψηφιότητες για την προσωρινή έδρα της αστυνομικής αδημίας σε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποχωρήσει από τον Μπράμσχιλ στο άτυπο συμβούλιο που έγινε στο Βίλνιο τον Ιούλιο φέτος υπευλήθησαν οι υποψηφιότητες των κρατών μαλλών και ζητήσαμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τη δυνατότητα πρόσβασης ε, στις διάφορες τοποθεσίες, ε, τη δυνατότητα ασυλίας ε, του προσωπικού, το να υπάρχει κατάλληλες εγκαταστάσεις, σχολεία για τα παιδιά των υπαλλήλων και ούτε καθεξής, καθώς επίσης και κάποιες ενδεικτικές ημερομηνίες για το πότε θα είναι πλήρως ε, διαθέσιμες οι εγκαταστάσεις αυτές. Από εκεί και πέρα ε, ακολουθήσαμε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, ευρωπαϊκές αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας επιλογής η Προεδρία είχε ως βασικό στόχο τη διαφάνεια και φυσικά εκμεταλλεύτηκε και την προηγούμενη εμπειρία και πρακτικές σε αντίστοιχες διαδικασίες. Είδαμε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Καταλήξαν σε, Κατέληξαν σε συμφωνία οι υπουργοί, αλλά η διαδικασία απαιτεί νομοθετική πράξη για τη συνέχεια, προκειμένου να αλλάξει επισήμως η έδρα της ε, Αστυνομικής Ακαδημίας, διότι βάσει του άρθρου 4 της απόφασης σύστασης ε, της ΕΠΟΛ, αναφέρεται ρητά ότι προς το παρόν η έδρα ε, βρίσκεται στο Μπράνσχιλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν δύο εναλλακτικέ λύσεις. Η μία περίπτωση είναι να υποβάλει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια νέα απόφαση της ε, ε, Αστυνομικής Ακαδημίας στο εγγύς μέλλον και αυτό τη ζητήθηκε να κάνει στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Σωτερικών Υποθέσεων του Ιουνίου στο οποίο οι Υπουργοί απέκλεισαν το ενδεχόμενο συγχώνευσης ε, Europol-Sepol, ε, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται και στην ε, άποψη της Επιτροπής της δικής σας. θα μπορούσαμε να έχουμε μια νέα απόφαση υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί πριν από το τέλος του 2014. Να επισημάνω εδώ ότι μας πιέζει και ο πολιτικός κύκλος των πολιτικών εξελέξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε και ευρωεκλογέ και επομένως ε, θα πρέπει να δράσουμε γέρος. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε μια δεύτερη εναλλακτική λύση, θα πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία τουλάχιστον ε, του ενός τετάρτου των κρατών μελών. Προς το παρόν είναι 7 τα κράτη-μέλη, τα οποία βάσει του άρθρου 76 υποπαράγραφος Β της συνθήκης Και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, η Προεδρία αποφάσισε να ξεκινήσει την προετοιμασία προκειμένου να μπορέσει να εγκριθεί η νομοθετική πράξη ε, μέσω διαδικασίας συναπόφασης πριν το τέλος του 2014, λαμβάνοντας και πάλι υπόψη, όπως σας είπα, και το γεγονός ότι έχουμε ευρωεκλογέ. Που σημαίνει ότι από τον Απρίλιο του χρόνου θα έχουμε μπει σε προεκλογική εκστρατεία. Ε, χρειάζεται συμφωνία λοιπόν ε, για να ληφθεί απόφαση. Υπάρχει βέβαια ένα κοινό συμφέρον, μας ενδιαφέρει να παραμείνει η ΣΕΠΟΛ σε λειτουργία και να μην μείνει το προσωπικό για πολύ μεγάλο διάστημα σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Τι μελιγενέστε τώρα. Εδώ τονίζουμε ότι η Προεδρία είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές ε, εγκαίρως και αυτά από πλευράς μου σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ξεκινήσει η συζήτηση με τα μέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων διευκρίνησε ότι η πρόταση για τη συγχώνευση Europol-Sipol παραμένει στο τραπέζι ως η μόνη λύση για τη συζήτηση. Σημειώθηκε ότι στην ε, συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο Συμβούλιο οι Υπουργοί κατέληξαν σε μια πολιτική απόφαση για μια προσωρινή έδρα της ΕΠΟΛ μετά από μια συνήθιστη διαδικασία και αυτό φυσικά είναι συνέπεια της ανακοίνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν μπορεί άλλο να φιλοξενεί ε, της Apple στο Bramshill στο μέλλον. Να σας υπενθυμίσω ότι το πεδίο εφαρμογής της πρότασής μας ε, είναι να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τρόπους να έχουμε αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία και κατάρτιση και αυτό γίνεται μέσω της μεταρρύθμισης της Europol με μια σειρά από επιχειρησιακές βελτιώσεις οι οποίες ε, Επίσης άπτονται και τις συνεργασίες ε, της Europol και τις συνέχισης δραστηριοτήτων οι οποίες γίνονται προς το παρόν από άλλες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και της Apple. Προσπαθούμε να έχουμε έναν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό ε, τρόπο και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και στην πρότασή μου ας ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε και τη συγχώνευση Europol-Sepol. Αυτή η απόφαση υπαγορεύτηκε από το στόχο να έχουμε συνέργεια και εξοικονόμηση πόρων, ε, καθώς και το συνολικό στόχο να μεταρρυθμίσουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία στη λεγόμενη κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ε, την οποία έχουν εγκρίνει και τα τρία θεσμικά όργανα. Συνεπώς, η θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο για να, θεωρεί, ε, να εξετάσει μεμονωμένα το θέμα αυτής της προσωρινής ε, έδρας θεωρούμε ότι είναι αμφίσιμο και αμφίβολο από πολιτικής και τεχνικής σκοπιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές ενστάσεις και από πλευρά Συμβουλίου και από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη δυνατότητα συγχώνευσης Europol-Sepol αλλά υπάρχουν και κάποιες φωνές υποστήριξης, ε, κυρίως ε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, σημειώνει με ικανοποίηση ότι γίνεται επικοδομητική πρόοδος και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις άλλες ε, πτυχές της πρότασής μας για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της Europol και ακριβώς αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της επιχειρησιακής και λειτουργικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της ΣΥΠΟΛ και της έδρας της. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία λύση η οποία θα προσπαθεί να εκλογικεύσει και να βελτιώσει τα πράγματα και να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους που σας ανέφερα προηγουμένως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, εσείς είστε υπέρ της συγχώνευσης Europol-Sepol ε, και θέλει να λάβει και ο κύριος Δίας Δεμέρα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Πρώτον, να εκφράσω το σεβασμένο μου στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, του Συμβουλίου. Οι επικρίσεις μου δεν είναι κατά της Προεδρίας του Συμβουλίου, είναι κατά του Συμβουλίου. Απορρίπτω κύριε Πρόεδρε τις εξηγήσεις που μας έδωσε σήμερα το πρωί η Προεδρία. Τις απορρίπτω και επί της ουσίας και επί της διαδικασίας. Και τις απορρίπτω διότι καταρχάς είναι εκπρόθεσμες. Αυτές οι εξηγήσεις έπρεπε να είχαν δοθεί εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πριν από τις 8 Οκτωβρίου. Επιπλέον τις απορρίπτω διότι είναι ανακριβείς. Διότι τους ενδιαφέρει η δική τους ερμηνεία της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά άρθρα και επίσης θεωρώ ότι είναι αδικαιολόγητες. Απορρίπτω επίσης ε, την πρόταση που αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει εφαρμοστεί καταλήλως το άρθρο 76β της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εφαρμοστεί σωστά το άρθρο 76β θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του Κοινοβουλίου πριν από τις 8 Οκτωβρίου, όχι σήμερα. Δεν εφαρμόστηκε σωστά λοιπόν και το άρθρο 294 το οποίο αναφέρεται στην νομοθετική ισότητα. Πολλοί γνωρίζουν και εγώ ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η ε, όμορφη πρωτεύουσα της αδελφού χώρας της Πορτογαλίας, αλλά πέραν αυτού η Λισαβόνα είναι η συνθήκη η οποία χωρεί εξουσία, εξουσία ε, αντίστοιχη με το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο. Δεν γνωρίζετε λοιπόν τι σημαίνει η συνθήκη της Λισαβόνας ή την ε, αγνοείτε τεχνιέντος. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω το εξής. Γίνεται μία ε, πρόσκληση χωρίς να μιλήσουν μαζί σας κύριε Πρόεδρε, χωρίς να μιλήσουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς να ενημερώσουν εμένα που είμαι ο αρμόδιος εισηγητής και όλα αυτά γίνονται μονομερός, γίνονται όλα στη σκιά, στο παρασκήνιο και όπως είπατε και εσείς υποβάλλονται 7 προτάσεις κύριε Πρόεδρε και εδώ μας έρχεται μία το Κοινοβούλιο δεν έχει αποφασίσει για αυτές τις 7 προτάσεις για τη νέα έδρα. Δεν μίλησε για την αγαπημένη μου Άβυλα. Ούτε για τη Ρώμη. Ή τη Χάγη. Ένα άλλο χτύπημα κάτω από τη ζώνη στα όσα ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε για το Τάμπερα. Ούτε για τη Βουδαπέστη, ούτε για τη Βέρεια, ούτε για το Λέμπρεμορ δεν έχει πει την άποψή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πει την άποψή του και δικαίω. Υπευλήθησαν λοιπόν οι προτάσεις, τις είδα και πραγματικά ντρέπομαι να το σχολιάσω. Είναι επονίδιστο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αλλά και τίποτα λιγότερο. Στι 8 του μηνό στο Λουξεμβούργο φτάσαμε πλέον στον κολοφόνα τη δόξα του, διότι χρησιμοποίησαν ένα μηχανισμό που μόλι μα εξήγησε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αμφίβολο το λιγότερο. Και από νομική πλευρά και από πολιτική πλευρά είναι αμφισβητήσιμη αυτή η διαδικασία, διότι εμεί είμαστε ένα πολιτικό κοινοβούλιο, πάρα πολύ πολιτικό κοινοβούλιο δεν έχει ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία και φυσικά επειδή δεν έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία το αποτέλεσμα είναι παράνομο. Και επιπλέον αντικειμενικά και μόνον και με όρος αριστείας έχω και εγώ τη δική μου την υποψηφιότητα και ξαφνικά έρχεστε εδώ για να μας φέρετε πρωτετελωσμένο. Και με μια επίφαση νομιμότητας αλλά δεν υπάρχει καμία νομιμότητα εδώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο επιζητά διαφάνεια, ζητά δημοσιοποίηση των στοιχείων και το Κοινοβούλιο ζητά να συμμετέχει ως συνομοθέτης όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και θέλει να πει την απόψή του αιτιολογημένα για κάθε μία από τις έδρες οι οποίες έχουν υποβληθεί ως πρόταση. Το πρόσχημα της προσωρινής έδρας είναι απλώς και, ένα και μόνο ένα πρόσχημα για να γίνει κάτι μόνιμο. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και το θέμα είναι τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι κατεπήγον και επομένω δεν είναι τελείως δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη αυτή η προσωρινή κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε απορρίπτω τρεις την πρόταση και απαιτώ να εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται από τη συνθήκη τη Λισαβόνας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Η κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιστώνω ότι ακόμα βρισκόμαστε σε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτή τη συγχώνευση, την οποία αρνούνται. Και ακούσαμε ότι σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες εδώ πρέπει να αποφασίσουμε εμείς είμαστε οι κυρίως αρμόδιοι αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να γίνει η συγχώνευση σε Πολ και Europol. Άκουσαμε άλλες επιτροπές να αποφαίνονται, αλλά τέλος πάντων οι άλλοι δεν έχουν αρμοδιότητα για το ναι ή το όχι των δύο αυτών υπηρεσιών της συγγόνωσης. Κύριε Πριμπέ. Θα πρέπει να δούμε ότι ανέλαβε κάποια πρωτοβουλία με υπευθυνότητα η Προεδρία για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, γιατί όπως και εσείς ε, υπενθυμίσατε, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει στο, στο να κλείσει το κέντρο και να πουλήσει εγκαταστάσεις, οπότε πια δεν θα έχει έδρα η ΣΕΠΟΛ. Οπότε θα πρέπει να βγούμε αυτό το διέξοδο και η Επιτροπή ε, έχει το, το, το, τα σχεδιά της, είναι κοινό μυστικό, το τι θέλει να κάνει. Το πρόβλημα δεν είναι η διαδικασία η οποία ε, επιδέχεται προς αμφισβητήσεις, αλλά το θέμα είναι ε, πάμε να, γίνει αυτή η συνάντηση 27 Νοεμβρίου για να φασίσουμε και θα πρέπει να δούμε σε εκείνη την ακρόαση πώς θα έρθουν οι εκπρόσωποι των 7 υποψηφίων χωρών για να μας παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Οπότε, εκεί 5-10 λεπτά ο καθένας να παρουσιάσει την πρότασή του. Να ακούσουμε τι έχει να πει η Ουγγαρία, η Ισπανία, η Ελλάδα και οι άλλοι. Οπότε, να έχουμε κάποια ιδέα εδώ στην Επιτροπή μας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προσφέρει κάθε χώρα. Δεν ξέρω τι λέει το Συμβούλιο, αλλά έτσι νομίζω μπορούμε στην Επιτροπή μας να αποφασίζουμε. Είπατε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση μέχρι το τέλος του έτους. Ε, έχετε όμως στο μυαλό σας και ένα καταρχήν ε, χρονοδιάγραμμα. Τι έχει να πει σχετικά με αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, πριν αυτό που είπατε. στήσεις Το, μεσημέρι, το μεσημέρι σήμερα θα το συζητήσουν οι συντονιστές. Θα προσεστούν εκεί οι προτάσεις και θα συζητηθούν. Οπότε και θα κρυφτεί το θέμα αυτή τη ακρόαση και κάθε υποψηφία πόλη θα προσθέσει εκεί τι προτάσει τη. Αυτό και θα συζητήσουμε τότε. Ο κύριο Κέρχοπ έχει ζητήσει όμω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω να πω τα εξή. Απεφάσισε το Ηνωμένο Βασίλειο να κλείσει τι εγκαταστάσει στο Μπράμσιλ. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, υπήρχαν προβλήματα οικονομικά. Άρα πρέπει να μετακομίσει η ΣΥΠΟΛ. Και εγώ δεν θέλω να γίνει η συγχώνευση των δύο υπηρεσιών, ΣΥΠΟΛ και Γύροπολ. Μια που ο ρόλος είναι διαφορετικός πέραν του τι θα αποφασίσει η Επιτροπή και πέραν του τι αρμοδιότητα θα έχει στο μέλλον η ΣΥΠΟΛ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αρμοδιότητες που θα προσδώσουμε στην υπηρεσία αυτή. Γιατί έχουμε τις ε, εθνικές διοκτικές αρχές, οι οποίες ήδη ασχολούνται με παρόμοια θέματα, αλλά να μην έχουμε επικάλυψη αρμοδιοτήτων και σύγχυση. Κάποια στιγμή θα αποφασιστεί αυτό τώρα όσον αφορά το πού θα μετακομίσει η σχολή. Εμεί είχαμε πει ότι είμαστε υπέρ του να πάει στις κάτω χώρες. Τώρα όμως έχουμε συγκεκριμένες υποψηφιότητες συγκεκριμένων πόλεων και το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συναπόφασης θα πρέπει να εξετάσει την διαθεμία που θες της υποψηφιότητας. Άλλαξαν πολλά με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά δεν θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, σε κοινοβουλευτική επιτροπή να μας έχουν ζητήσει να αποφανθούμε για την έδρα κοινοτικού θεσμικού οργάνου. Έχουμε ισορροπία δυνάμεων, με διάφορες πιέσεις, θα πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή. Γι' αυτό θα πρέπει να κατησχύσει σαν κριτήριο και όχι το αν είναι πιο ελκυστικό ένα μέρος από άλλο. Και γι' αυτό σας λέω, δεν έχω καμία ένσταση να πάει η σχολή στη Βουδαπέστη. Και δεν ξέρω αν διαδικασία που έχουμε αποφασίσει αν είναι πιο σωστή και αν θα είναι αποδεκτή από τα άλλα θεσμικά όργανα. Άρα, εμεί που και πάρα πολύ χρόνο πάνω σε αυτό, αλλά θα πρέπει τέλο πάντων να αποφασιστούν ποιε θα είναι οι λειτουργίε τη ε, ΣΥΠΟΛ. Και από την άλλη μεριά να δούμε και πού θα εγκατασταθεί στο μέλλον αυτή η υπηρεσία. Ευχαριστούμε κύριε Κυριακόπουλο. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω στα ουγγρικά ωστόσο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και το ίδιο το Κοινοβούλιο κατ' επανάληψη έχουν τονίσει ότι είναι κατά της συγχώνευσης Ευρωπόλ και ΣΕΠΟΛ. Έχουμε τονίσει μάλιστα ότι θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουν ανεξάρτητες οι δύο αυτές οργανώσεις, οι δύο αυτοί οργανισμοί καλύτερα. Τώρα, πώς θα διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία αυτή, αρχίζει και γίνεται αντικείμενο διαθεσμικής, διοργανικής συζήτησης. Πρέπει να βρούμε λοιπόν κάποιο κοινό έδαφος ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η κατάσταση φαίνεται πάντως ε, να γίνεται ενδιαφέρουσα διότι το Κοινοβούλιο μέχρι τώρα ποτέ δεν είχε τη δυνατότητα να εγκρίνει μόνο του τις έδρες ε, των οργανισμών ή να λαμβάνει υπόψη του οικονομικές παραμέτρους για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. Δεν ε, νομίζω λοιπόν ότι έχουμε δικαίωμα να επικρίνουμε το Συμβούλιο και εν πάση περιπτώσει μια διαδικασία η οποία πάντοτε διεξήχθη με τον ίδιο τρόπο, όπως και τώρα δηλαδή. Το Συμβούλιο μάλιστα υπήρξε ομόφωνο και αυτό νομίζω ότι ο λόγος δηλαδή για την ομοφωνία αυτή του Συμβουλίου είναι λόγω της ποιότητας της Ουγγρικής προτάσεως. Δεν είναι δική μας δουλειά να επικρίνουμε το Συμβούλιο για τις επιμέρους αποφάσεις που λαμβάνει ε, για τις προτάσεις που κάνει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε τη συγκεκριμένη αυτή απόφαση. Είμαι βέβαια ότι το Συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση διότι πιστεύουν, πιστεύουν οι Υπουργοί δηλαδή, ότι όντως η Ουγγρική πρόταση είναι οι καλύτεροι. Πρέπει να εξετάσουμε βέβαια το διαθεσμικό πρόβλημα, ώστε να είναι και τα δύο θεσμικά όργανα ικανοποιημένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις διευκρινήσεις που άκουσα ως τώρα από Κομισιόν Συμβούλιο και από τον εισηγητή μας τη Μέρα. Εγώ που είμαι όμως και για την Ευρωπόλ και την ενδεχόμενη συγχώνευση με τη ΣΕΠΟΛ, έχω κάποιες ερωτήσεις και έχω και ένα σχόλιο, γιατί είμαι και εισηγητής για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέματα μάλιστα τέτοια έχουν θίξει και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Ουγγρικής κυβερνήσεως. Η δική μου ερώτηση είναι, εάν υπό το φως τώρα της εκθέσεως της Ευρωπόλ που περιέλαβε στην πρόταση της Κομισιόν, πρόταση συγχωνεύσεως δηλαδή, και εγώ και η ομάδα μου, ήμασταν πάντοτε κατά της συγχώνευσης που θα μετέφερε βέβαια στην περίπτωση αυτή το αρχηγείο της ΕΠΟΛ στην Χάγη. Διερωτώ με αν δεν χρειαζόμαστε νέα πρόταση της Κομισιόν για νέα διαδικασία συναπόφασης το οποίο θα καθορίσει κιόλα πώ θα εργαστούμε εδώ στην Επιτροπή μα. Διότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε την έκθεση Ντεμέρα, μετά να προχωρήσουμε σε τριμερή διάλογο και συναπόφαση με το Συμβούλιο, πριν να εξαντλήσουμε το εάν το θέμα δηλαδή, αν θα απορρίψουμε την συγχώνευση Ευρωπόλ και ΣΕΠΟΛ. Πρέπει δηλαδή πρώτα να κλείσουμε την μία νομική, νομοθετική διαδικασία πριν να αρχίσουμε νέα. Οπότε τότε θα χρειαζόμαστε και νέα έκθεση. Θέλω λοιπόν να επιβεβαιώσω και από άποψη προθεσμιών. Τι πιστεύετε κύριε Πρόεδρε ότι μπορεί να γίνει με τη διαδικασία αυτή αν δηλαδή όντως μπορούμε να τηρήσουμε την προθεσμία του τέλους του 2014 που θα ήθελε να τηρηθεί και το Συμβούλιο. Τώρα, διακόπτει ο Πρόεδρος. Έχουμε κάπως περάσει το χρόνο μας και έχουμε και ηλεκτρονική ψηφοφορία σε λίγο. Αν είναι δυνατόν λοιπόν να επιταχύνουμε λίγο τις παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σταβάρης. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, η δική μου θέση ως εισηγητού για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία θέλω να διευκρινίσω το εξή. Όχι μόνο δεν έχω ένσταση για την Βουδαπέστη ως αρχηγείο της ΣΕΠΟΛ, μάλιστα συγχαίρω τη Βουδαπέστη για την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα κατά προτεραιότητα θέματα για το Κοινοβούλιο, δηλαδή κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. θα ε, συζητηθούν επαρκώς. Αναμένω από το Κοινοβούλιο να είναι συνεπές με τη θέση του ιδίως δηλαδή εάν πρόκειται να έχουμε εξουσίες συναπόφασης για το θέμα. Και ελπίζω επίσης το γεγονός ότι η απόφαση αυτή έχει τεθεί επιτάπητος θα οδηγήσει και σε επιτάχυνση της διαδικασίας για την ψήφιση του ψηφίσματος. Αυτά θέλω λοιπόν από για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ που είμαι σκιώδης συγκίτρια για μη υπάρχουν θέμα που είναι το θέμα της ΕΠΟΛ, εγώ θέλω να πω ότι είμαι ευγνώμων, ιδιαίτερα ευγνώμων στο Συμβούλιο, διότι έλαβε αυτή την ανεπίσημη απόφαση. Βεβαίως ε, δεν είναι επίσημη. Η Κομισιόν γνωρίζει ακριβώς την θέση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την συγχώνευση Ευρωπόλ και ΣΕΠΟΛ. Εμείς μάλιστα έχουμε ζητήσει ε, με επίταση από την Κομισιόν να προχωρήσει, γιατί πρέπει να βρεθεί βεβαίως αρχηγείο για την ΣΕΠΟΛ και να δοθεί και τελική μορφή στην έκθεση αυτή. Βέβαια και το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει και ελπίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία είτε προς τη μια κατεύθυνση είτε προς την άλλη πριν από το τέλος της θητείας μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα υπησέλθω τώρα στις λεπτομέρειες ε, των επιχειρημάτων κατά της συγχωνεύσεως, γιατί τα έχουμε πολλές φορές εδώ. Μόνο θα πω ότι εάν συζητούμε τις διάφορες πτυχές της κίνησης αυτής για την εξέβρεση νέου αρχηγείου, πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά πόσον αυτό θα εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της ΣΕΠΟΛ, κάτι που θεωρούμε άκρας σημασίας και από την άλλη μεριά έχει ληφθεί απόφαση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι όταν αναζητούμε νέες έδρες για ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προτεραιότητα δίνεται στις νέες χώρες μέλη. Ουγγαρία και Βουδαπέστη, από όσο γνωρίζω στην περίσταση αυτή, ήταν η μοναδική πρόταση που προερχόταν από νέα χώρα μέλος. Και αυτό ήταν και ένα επιχείρημα υπέρ της πρότασης αυτής. Τώρα, για να έρθω λίγο σε ορισμένες από τις ανησυχίες που ακούστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ιστορικό της ε, Ουγγρικής κυβερνήσεως. Ελπίζω ότι μέχρι ότου να φτάσει να μετακομίσει σε πόλ, η Ουγγαρία θα έχει νέα κυβέρνηση. Θα γίνει αυτό σίγουρα το επόμενο χρόνο, τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το πρώτο εξάμεινο του επόμενου χρόνου. Και είμαι βεβαία ότι η επόμενη κυβέρνηση θα έχει πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερη απόδοση σε θέματα κράτους δικαίου και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Άρα το επιχείρημα αυτό θα εκλείψει. Τώρα, σχόλια για την πολιτική συζήτηση. Νομίζω ναι, είναι σημαντικό να μην αχθεί σε πολιτικό επίπεδο, γιατί δεν απαραίτητα πολιτική συζήτηση. Αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες στην Ουγγρική Βουλή, το κόμμα Φίντες έστρεψε το θέμα αυτό σε πολιτικό θέμα. Και η MSP αποκλήθηκε από το για η αντιπολίτευση δηλαδή, προδότες. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα αυτά τα πράγματα να τα αποφύγουμε τέτοιες πολιτικές αντιπαραθέσεις και να αφήσουμε την Βουδαπέστη να έχει τις πιθανότητες να επιλεγεί ως έδρα για την ε, ε, Βλέπω ότι έχετε ένα σχόλιο ακόμα κύριε Ντεμέρα γιατί κάπως έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο σκέψεις. Η συνήθις νομοθετική διαδικασία που ακολούθησε ε, το Συμβούλιο θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στο νομικό κριτήριο της ε, σταθμισμένης πλειοψηφίας. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι αμφισβητήσιμος ο μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιήθηκε με βάση κατά αποκλεισμό διαδικασία. Αρχικώς η Φιλανδία και η Ελλάδα αποκλείστηκαν, μετά η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά πριν από αυτό η Φιλανδία πέσυρε την υποψηφιότητά της για να υποστηρίξει δημοσίως ε, την κάτω χώρες. Αυτή η διαδικασία είναι τουλάχιστον παράτυπη και αμφίβολη. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απαντήσω στους συναδέλφους. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέει η Βερονίκ. Έχει πολύ λογική αυτό που ακούσαμε το να υπάρχει απαραίτητη συμμετοχή και η νομοθετική ε, ε, διαδικασία να ακολουθηθεί με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητηθεί το Νοέμβριο το θέμα για να μπορέσουν να έρθουν οι υποψήφιες χώρες να μας παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους. Για αυτά που λέει ο συνάδελφο Τίμωθη Κίρκοπ. Και εγώ συμφωνώ μαζί σα, Δεν θέλω τη συγχώνευση. Απορρίπτω αυτή τη συγχώνευση Ευρωπόλ-ΣΕΠΟΛ υπέβαλα 122 τροπολογίες στην νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ λοιπόν ότι οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση και μάλιστα με το ίδιο σκάφος. Σίγουρα πρέπει να μερετήσουμε όλες τις έδρες, όπως λέει η Βερονίκ, και βεβαίως διαφωνώ και με την ε, ιδέα αυτής της κατανομής, διότι αυτή είναι αντίθετη στην ε, ε, ιδέα της αριστείας. δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μια, ένα καταμερισμό ο οποίος θα μας οδηγήσει σε χειρότερη έδρα όταν θα μπορούμε να έχουμε την καλύτερη. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Στη συνάδελφο Κίνγκα Γκάλ. Με όλο το σεβασμό Κίνγκα εξακολουθώ να είμαι υπέρ του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι το πρώτο τμήμα της παρέμβασης του κυρίου Ταβάρες, ε, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε ένα ε, σχόλιο για την Κίνγκα Γκάλ, τη συνάδελφα από την Ουγγαρία. Κοίταξε να δεις Κίνγκα και έχω εδώ την κατανομή των ε, αποκεντρωμένων οργανισμών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει Ουγγαρία οργανισμό, αλλά δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Κύριε Πρόεδρε, να πω το εξή. Είναι ψευδέ το επιχείρημα του κατεπήγοντα χαρακτήρα. Και γιατί αυτό, διότι η έδρα του Μπράμσχιλ είναι χωρισμένη στη μέση. Το ένα τμήμα ανήκει στη ΣΕΠΟΛ και το άλλο τμήμα στη Βρετανική αστυνομία. Για να απολυθεί το κτίριο, το μας είπαν ότι ο χρονικός ορίζοντας της πώληση είναι ε, Μάρτιος Άνοιξη του 2014. Αλλά η ε, Βρετανική αστυνομία θα μπορεί να μείνει μέχρι το 2015, ένα χρόνο αργότερα. Είναι λογικό ότι αν το εκχωρήσουν στην αστυνομία, επειδή δεν θα μπορέσουν να το πουλήσουν, θα μπορούν να το εκχωρήσουν και στη Ευρωπαϊκό, στην ε, ΣΕΠΟΛ. Είναι λοιπόν ψευδές αυτό το επιχείρημα ότι είναι πήγον να βρούμε μια νέα έδρα. Επίσης, η Επίτροπος έγραψε επιστολή στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να τους πούνε επακριβώς πότε θα πρέπει να ε, αποχωρήσει η ΣΕΠΟΛ από το κτίριο του Μπράμσχιλ. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία μόλις ξεκίνησε κύριε Πρόεδρε και θα πρέπει να συνεχίσουμε με το ρόλο που εκχωρείται σε θέματα συναπόφασης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε κύριε Διαστεμίρα. Ε, ακούσαμε την πρόταση του συντονιστή του ΕΛΚ, ε, ακούσαμε και την κυρία Βερονίκ Ματιέ για την ακρόαση για να έρθουν όλοι οι εκπρόσωποι από όλες τις έδρες θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό στη συνεδρίαση των συντονιστών. 27 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που προτείνεται ως πιθανή για την ακρόαση. Ε, θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα και τώρα όμως πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο διότι πρέπει να ψηφίσουμε στις 10.30 και έχουμε ένα ακόμα θέμα να συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Παπα-Νικολάου για τη ε, διαχείριση των επιστροφών, συνεργασία με τρίτες χώρες, αποτελεσματική εφαρμογή συμφωνιών και πρακτική εφαρμογή τη οδηγίας περί της επιστροφής. Πρόκειται για το σημείο υπαριθμών 6 της ημερήσιας διάταξης. Προτείνω λοιπόν να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων εδώ να ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή μας, τον κύριο Παπα-Νικολάου. Μετά θα ε, μιλήσουμε για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, την προθεσμία κατάσταση τροπολογιών κλπ. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας εδώ η οποία έφτασε στην Επιτροπή μας μετά από τη συζήτηση που έγινε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Τίτλος είναι «Διαχείριση της επιστροφής, συνεργασία με τρίτες χώρες, αποτελεσματική εφαρμογή συμφωνιών και πρακτική εφαρμογή της οδηγίας περί της επιστροφής». Πρόκειται για συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων και όταν έγινε η πρόταση από το ΕΛΚ, ο αρχικός τίτλος ε, ήταν για να συζητήσουμε τις ελλείψεις που έχουμε και την έλλειψη ε, ενός συνολικού ε, συστήματος για τις επιστροφές. Να σας πω το σκεπτικό μας. Έχουμε ένα κοινό σύστημα σύλλου, έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση εντός εισαγωγικών για το κοινό σύστημα διαχείρισης συνόρων και κατά την άποψή μας, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά αυτά τα συστήματα, θα πρέπει να υπάρχει και ένα συνολικό ε, σύστημα διαχείρισης των, ε, της μετανάστευσης. Και θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο αν υπήρχε και ε, συμφωνία και κατάλληλος καταμερισμός μεταξύ των κρατών μαλλών για ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Και να σας διευκρινίσω ευθύς εξ αρχής ότι όταν αναφερόμαστε στις επιστροφές δεν αναφερόμαστε σε τούντες άσυλο οι οποίοι μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο αν επιστραφούν στη χώρα καταγωγής τους και αυτό το διευκρινίζω ευθύς εξ αρχής. Χρειαζόμαστε μια συνολική πολιτική μετανάστευση και η πολιτική για τις επιστροφές είναι υψής της σημασίας στον τομέα αυτό. Αναφερόμαστε λοιπόν στους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι ε, αυτή τη στιγμή έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που τους παρέχει το σύστημα ασύλου και τις ε, διαδικασίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και τους έχει αρνηθεί η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν ε, πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να επιστραφούν στις χώρες τους. Γίνονται σεβαστά πλήρως τα δικαιώματά τους και υποστηρίζονται και από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Βέβαια πρέπει να υπάρχει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για το θέμα αυτό, διότι είναι περίπλοκο. Και εγώ από την αρχή ήμουνα ιδιαίτερα θετικός ε, για την ε, αλλαγή του τίτλου και θα ξαναφερθώ σε αυτό και ε, εδώ αναφέρεται στον τίτλο και η οδηγία περί της επιστροφής και ελπίζω ότι όλες οι ομάδες θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κοινά συμπεράσματα ακριβώς λόγω αυτού του συμβιβασμού. Ε, υπάρχουν πολιτικές διαφορές ε, σε αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα, αλλά φρονώ ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συνολικό πρόγραμμα για τις επιστροφές, ε, μια συλλογική προσέγγιση για την διαχείριση των επιστροφών και να δώσουμε ιδέες και να συνεισφέρουμε στην διοργανική συζήτηση που γίνεται για το όλο θέμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τμηματική προσέγγιση και οι προσεγγίσεις μας είναι εντελώς κατακαιρματισμένες και υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα κυρίως στο νότο και στα νοτιοανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι γίνεται με τις πολιτικές για τις επιστροφές και θέλουμε και συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δείτε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 για τη Συμφωνία για τις Επιστροφές, ένα βασικό στοιχείο της έκθεσης αυτής είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και στοιχεία. Η έκθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Είμαστε στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας και στο τέλος της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά και στο τέλος του προγράμματος της Στοκχόλμης και εγκριθεί και το νέο πολιτές ε, πρόγραμμα για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Θα παρουσιαστεί από ό,τι είδα στο χρονοδιάχρημα λίγο πριν ε, την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία για τις επιστροφές και θα ψηφιστεί ε, λίγο μετά. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστική. Υπάρχει και η τραγωδία στη Λαμπεντούζα. Όλα όσα συνέβησαν την περασμένη Δευτέρα στην Ελλάδα ε, διεσώθησαν 75 μετανάστες ε, στη θάλασσα στην Ελλάδα και έχουμε και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλη εισρωή μεταναστών στην περιοχή της Μεσογείου και οι χώρες της ε, Νοτιού Ευρώπης ε, κυρίως είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εισαγωγικά και από εκεί και πέρα μπορώ να ακούσω σχόλια και προτάσεις από τους κοιόδης εισηγητές, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων, όπως επίσης και όλους τους συναδέλφους σε όλες τις πολιτικές ομάδες, διότι είμαστε ανοιχτοί προ συζήτηση, προτάσεις, ε, οτιδήποτε έχετε τις επόμενες εβδομάδες. Καταρχάς, η αρχή της ε, μη επαναπροώθησης θα πρέπει να γίνεται πάντα σεβαστή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι υψής της σημασίας για όλους μας και φυσικά όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφαρμογή των διμερών συμφωνιών. Δεύτερον, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και των ευρωπαϊκών και των διμερών ε, συμφωνιών επιστροφών. Υπάρχουν στοιχεία για την εφαρμογή των συμφωνιών επιστροφών. Το Κοινοβούλιο ανέλαβε να συντάξει αυτή την έκθεση και ζητά και σήμερα ε, και πρέπει να λάβει αυτά τα στοιχεία. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσο θα μας δοθούν. Και επίσης υπάρχουν διμερείς συμφωνίες ε, στις οποίες δεν έχουμε σχεδόν καθόλου στοιχεία. Και αν υπήρχαν τα στοιχεία αυτά, θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια αξιολόγηση για να δούμε τι έχει αποτέλεσμα και τι δεν έχει. Ε, έχουμε κάποια στοιχεία που μας δείχνουν ότι οι διμερείς συμφωνίες σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται καταλήλως. Το αυτό ισχύει και στις ευρωπαϊκές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Το καλύτερο παράδειγμα νομίζω είναι το Πακιστάν που έχω να σας περιγράψω. Η συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Πακιστάν Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λεπτομερή στοιχεία για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών ε, ε, Επανεισδοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς έχει ακριβώς η κατάσταση για τη συνολική εικόνα που έχουμε και τι στοιχεία <coughs> αριθμητικά έχουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τρίτον, η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ε, να ασχοληθεί περισσότερο με τα θέματα της διαχείρισης των επιστροφών. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτό στην ε, πολιτική της ε, ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης. Υπάρχει και μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανάπτυξης για το θέμα αυτό και νομίζω ότι ε, θα το αναφέρει αυτό και η Επιτροπή Ανάπτυξης. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητηθούν αυτά τα θέματα, όχι με την Επιτροπό Μάλστρομ μόνο, αλλά και με την Κάθριν Άστον και ίσως και με τον κύριο Φανορόμπαϊ ή οποιονδήποτε θα αναλάβει τα ενία στο μέλλον. Τέταρτον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, προτιμούμε τις εθελοντικές επιστροφές. Να καθορίσουμε ε, Ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ και να ευνοήσουμε αυτέ τι μορφέ επιστροφών. Επίση να πω ότι υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλιο για το θέμα αυτό μέχρι το 2014. Τώρα κάποια κονδύλια συγχωνεύονται, αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική δράση για τα κράτη-μέλη. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά και πάλι οι εθελούσιε επιστροφέ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πολιτική μας για τη διαχείριση των επιστροφών. Και τέλος θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες και θα πρέπει να εξετάσουμε την ευρύτερη εικόνα προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο, να δούμε τι γίνεται με την παράνομη μετανάστευση, να δούμε τους ε, ε, παράνομους μετανάστες, ε, το τι γίνεται με το λαθρεμπόριο και την εμπορία ανθρώπων και φυσικά να δούμε και τι γίνεται με τις χώρες διέλευσης, τις χώρες transit θα πρέπει να εντείνουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για τους λαθρεμπόρους οι οποίοι συλλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο και αυτό αποτελεί προτεραιότητα διότι θα πρέπει να ζητήσουμε προληπτική δράση στον τομέα αυτό και στον τομέα της, ε, του τράνζιτ. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις. Η συνεργασία δεν ξεκινά ούτε τελειώνει στο σημείο της επιστροφής. Θα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει κονδύλια σε τρίτες χώρες για την ε, βελτίωση των υποδομών τους και της οικονομίας τους και αυτό φυσικά θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γι' αυτό θα θέλαμε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης και αυτοί θα δώσουν την ε, συνεισφορά τους στο θέμα αυτό και θα πρέπει και οι τρίτες χώρες να προσπαθήσουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, ολοκληρώνοντας, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή, ότι δεν μα αρέσει η διαδικασία των επιστροφών και δεν θα θέλαμε στην πραγματικότητα να επιστρέφει κανεί. Θα θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο να είναι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε ένα συλλογικό σχέδιο και μια αποτελεσματική πολιτική μετανάστευσης. Αν δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, τότε δεν χρειαζόμαστε ούτε καν κανόνες ασύλου, ούτε χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Δεν θα πρέπει να γίνεται παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν θα πρέπει να επιστρέφει ένας παράνομος μετανάστης, ο οποίος έχει εξαντλήσει όλες τις ποθηνές νομικές δυνατότητες και καταχράται το σύστημα. Όταν υπάρχει κατάχρηση, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, πρέπει κάτι να γίνει ή μια τρίτη χώρα η οποία ζητά αναπτυξιακή βοήθεια για να μπορέσει να αναπτυχθεί ε, να μην ε, σέβεται τις υποχρεώσεις της. Κανείς δεν λέει ότι θα πρέπει να είναι τα πάντα τέλεια, αλλά υπάρχει ανάγκη να λιβάνονται κάποια μέτρα. Ε, δείτε την Τουρκία για παράδειγμα. Είναι μια χώρα η οποία λαμβάνει χρηματοοικονομική βοήθεια για να βοηθά τις ανθρώπους οι οποίοι περνούν από τη χώρα τους πώς μπορούμε να έχουμε χιλιάδες παράνομους μετανάστες οι οποίοι ταξιδεύουν στη χώρα και στα ευρωπαϊκά σύνορα. Ε, κύριε Παπα-Νικολάου, μπορείτε να ολοκληρώσετε, ναι, ένα λεπτό. Και να αφήνουμε τους λαθρεμπόρους να δρούν ανενόχλητοι, χωρίς να αναλαμβάνει δράση. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα. Δεν θα πρέπει να επιβληθούν ε, μέτρα σε τέτοιες τόσο προφανείς περιπτώσεις. Και επίσης να πω ότι κάποιοι λένε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ε, σύστημα εθελοντικής επανακατάστασης, γνωρίζετε ποια είναι η θέση μου επ' αυτού, για να υπάρχει αντίστοιχος καταμερισμός του βάρους μεταξύ κρατών μελών. Παρά το γεγονός ότι εγώ διαφωνώ και λέω ότι πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα τέτοιο σύστημα, ας δεχτούμε ότι δεν θα υπάρξει. θα μένουν οι άνθρωποι στην πρώτη χώρα στην οποία ε, φτάνουν, χωρίς να έχουν καμία ελπίδα για καλύτερο μέλλον, γιατί στις χώρες αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα απορροφησής τους. Υπάρχει πρώτη χώρα εισόδου, δεν υπάρχει επανεκατάσταση, δεν υπάρχουν επιστροφές. Οι κανόνες Σέγγεν δεν επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων αυτών σε άλλες χώρες. Εάν λοιπόν η κατάσταση μείνει έτσι, μακροπρόθεσμα, αντιλαμβάνεστε τι αποτελέσματα θα προκύψουν και τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι χώρες αυτές. Και ήδη αντιμετωπίζουν αυτό το διάστημα. Τα λέω όλα αυτά για να ε, βοηθήσω να ε, προληπτικά τα επιχειρήματα τα οποία θα παρουσιάσουν κάποιοι συνάδελφοι κατά των επιστροφών. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Υπάρχουν πολλά κοινά, ε, κενά, μεγάλη έλλειψη αποτελεσματικότητας. Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση και στην έκθεση, κατά την άποψή μα μπορούμε όλες οι πολιτικέ ομάδε μαζί να επισημάνουμε πολύ σημαντικά θέματα στα οποία συμφωνούμε. Κάτι τελευταίο, θα θέλαμε οι συζητήσεις αυτές ε, να οδηγήσουν ίσως σε κάποια συμπεράσματα. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας η οποία θέλει να συνεισφέρει στα προβλήματα και στα κενά που έχουμε. Το υπενθυμίζω την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε λίγο αυτή την πολιτική. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε κοινό έδαφος. Θέλω να ακούσω όλους τους σκιώδεις συζητητές ε, και θα συνεργαστώ καλή την πίστη με όλους και είμαι στη διάθεσή σας και σήμερα και στο εγγύης μέλλον για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να έχουμε ε, κοινά συμπεράσματα για τη ε, ε, διαχείριση των επιστροφών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γκυγιόμ, η κυρία Ρομέρο Λόπες και εάν ακόμη κάποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο παρακαλώ να το πράξει τώρα. Κύριος Ιακολίνο. Βλέπω και κανένα δυο χέρια ακόμη αλλά τότε περιοριστείτε στα δύο λεπτά γιατί 10 και 30 αρχίζει η ψηφοφορία. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ο λόγος και στην Κομισιόν και στην Προεδρία. Ε, να μην βρεθούμε σε δυσκολίες γιατί όπως είπα 10.30 και μισή αρχίζουμε. Η κυρία Γκυλιόμ. Είναι βέβαια πολύ επίκαιρα τα θέματα αυτά των επιστροφών. Επανέρχομαι στον τίτλο της ε, έκθεσης αυτής πρωτοβουλίας, διότι μιλούμε για συνεργασία με τρίτες χώρες, με εφαρμογή συμφωνιών και πρακτική εφαρμογή της οδηγής περί της επιστροφής. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ευρύτατο το θέμα. Ασφαλώς θα χρειαστεί να δουλέψουμε πάνω στους ορισμούς και σε μια πλαισίωση της προσέγγισης έτσι ώστε να είναι πιο ξεκάθαρα τα θέματα. Αυτό το πολυδιάστατο μπορεί να έχει αντικτυπώ και στο χρηματοδοτικό. Διότι μιλούμε τώρα για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, ο κ. παπα το γνωρίζει καλά και πρέπει να μην λησμονούμε ότι η προσέγγιση του Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη. Για το θέμα αυτό Υπάρχει προτεραιότητα η οποία δίνεται στην κοινοτική χρηματοδότηση στις εθελοντικές επιστροφές, στις εναλλακτικέ επιλογές για την κράτηση και ε, για το θέμα της ε, αναγκαστικής επιστροφής. Αλλά πρέπει να προωθούν σωστά οι προτεραιότητες. Για το πρώτο τμήμα της εκθέσεως που αναφέρεται σε συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες, έχω ορισμένα σχόλια εδώ. Θα τα δούμε βέβαια τα έθιξε και ο Γιώργος πριν από λίγο, να είναι σαφές ότι συνεχίζουμε να καταδικάζουμε τις αποκλήσεις στις ε, εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής. Ορισμένες χώρες μέλη εξακολουθούν να ε, εφαρμόζουν διμερείς συμφωνίες τις οποίες είχαν συνάψει πριν από την θέση ισχύ της κοινοτικής νομοθεσίας. Επίσης να συνεχίσουμε να καταγγείλουμε τον αδιαφανή χαρακτήρα ορισμένων συμφωνιών που έχει συνάψει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε δυσκολίες να βρούμε δεδομένα, έχουμε δυσκολία να τα χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε τις ε, συμφωνίες επιστροφής. Επίσης, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην εφαρμογή των συμφωνιών αυτών, είτε διμερών είτε κοινοτικών υπάρχει δυσκολία μέχρι και αδυναμία ε, των προσώπων να ε, βρουν να χώρο στη διαδικασία ασύλου και ούτε καθεξής. Τελευταίο στοιχείο για το τμήμα αυτό των ε, συμφωνιών επιστροφής χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία αυτού, αυτού του θέματος του μαστιγιού και καρότου για την εφαρμογή των συμφωνιών και πιο γενικά συνεργασία με τρίτες χώρες. Είναι αναγκαίο η πολιτική της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών να γίνει σε βάση ισορροπημένων και ξεκάθαρων προϋποθέσεων. Από τη μια μεριά η πολιτική των ε, επανεισδοχών επιστροφών και από την άλλη μεριά οι απειλούμενες κυρώσεις για τη μη εφαρμογή. Δεύτερο τώρα για την εφαρμογή της οδηγίας επιστροφής. Σημειώνω πρώτα ότι η Κομισιόν μέσα Δεκεμβρίου θα υποβάλει την πρώτη της έκθεση για την ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Δεν θα έχουμε μάλλον στοιχεία πριν από τη δημοσίευση αυτή της έκθεσης, ούτε και πριν από την ε, υποβολή των σχετικών τροπολογιών. Είναι λοιπόν σημαντικό να δώσει <coughs> τις πρώτες ενδείξεις η ε, Κομισιόν για το περιεχόμενο της έκθεσης, για να συμβάλλει έτσι στον προβληματισμό μας. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ορισμένες διατάξεις πρέπει να ε, μελετηθούν και ιδίως το θέμα της κράτησης, διότι έχει καταδειχθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις το μέτρο της κράτησης δεν ήταν το, το ίστατο μέτρο που ε- λήφθη, ενώ υπήρχαν άλλες εναλλακτικές επιλογές πιο πριν. Άρα θα έχουμε πολλή δουλειά και για να ξεκαθαρίσουμε τα προβλήματα και να δούμε τις ε, οικονομικές τους επιπτώσεις. κυρία Ρομέρα Λόπες, συγγνώμη. Μην τα λέτε εμένα κύριε Πρόεδρε όταν ο εισηγητής ε, μίλουσε 15 λεπτά. Κάπως πρέπει να κατανέμετε το χρόνο καλύτερα. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά κοιτάξτε, στις 10.30 έχουμε να ψηφίσουμε. Τα λαμβάνω όλα υπόψη. Σα παρακαλώ, κύριε Ρόμερο Λόπεθ. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Δεν υπάρχει όμω. Είναι ο εισηγητή, είναι ο εισηγητή, τονίζει ο πρόεδρο. Είναι φυσιολογικό να έχει περισσότερο χρόνο ο εισηγητή από ότι οι υπόλοιποι αγορητέ. Βοηθήστε να διαχειριστούμε τον χρόνο που έχουμε. Gracias, señor presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι επίγοντος χαρακτήρα αυτή η έκθεση, γιατί πρόκειται για κάποια οδηγία που αποτελεί ντροπή. Ε, το θέμα δεν είναι ότι είμαστε κατά των μεταναστών που έρχονται παράνομα και σε σχέση με την επιστροφή τους. Μακάρι να μην συνέτρεχε τέτοιος λόγος. Το θέμα είναι ότι είναι δυνατόν αυτοί να μείνουν μέχρι και έξι μήνες σε αυτά τα κέντρα όπου κρατούνται. Και αυτό αποτελεί παραβίαση των θεμελιδών του δικαιωμάτων. Αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί. Και αυτό το επιτρέπει η οδηγία μέχρι τους έξι μήνες. Και θα πρέπει επομένως να δούμε τι θα γίνει με τις μη κυβερνικές οργανώσεις γιατί έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια ε, κράτηση και φιλοξενίας όπου δεν έχουν πρόσβαση μη κυβερνήσει οργανώσει. Ασχολούνται μόνο οι διοικητικές αρχές. Δεν έχουν δικαιώματα. Θα πρέπει επομένω να βρεθούν οι μηχανισμοί για να τηρηθούν τα βασικά δικαιώματα. Και είναι δυνατόν να κάτσουν τρεις μέρες στην ε, Γερμανία και να υπάρχει εγγύηση τήρησης των θεμελιών δικαιωμάτων αλλά 20 τόσες μέρες στην ε, Ισπανία και 6 μήνες στην Ελλάδα καθυστερούν μέχρι να τους επιστρέψουν. Άρα θα πρέπει να βρεθούν οι μηχανισμοί για να κατοχυρωθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν μας είπε καμιά ημερομηνία η Επίτροπος, μάλιστα όπως το είπε η σύντροφος Σιλβιδρή, έχουμε κανένα στοιχείο. Έχουμε απλώς χιλιάδες πολιτών τρίτων χωρών που τώρα βρίσκονται σε κατάσταση που είναι αξιολύπητη. Οπότε μπορούμε να χαιρετήσω αυτή την εκθέση τη πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουμε με τρόπο, το ώστε να αλλάξει η κατάσταση που φερόμαστε σαν να είμαστε δουλέμποροι. Δεν φερόμαστε σαν να είμαστε Ευρωπαίοι μια Ευρώπη πολιτισμένη. ή αλλού. Επομένω, τηρούνται αλλά δεν τηρούνται καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό θα πρέπει άρδιν να αλλάξει. Euh, monsieur le Président, excusez-moi de râler comme d'habitude, mais en règle générale, vous donnez la parole au shadow rapporteur en premier, donc à un. Παραπονιέμαι και πάλι. Α, θα, θα πρέπει πρώτα να μιλάω ως και ο ένας για κάθε πολιτική ομάδα. Απαράδεκτη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ τον εισηγητή και θεωρώ ότι αν, αν με άκουγε θα ήταν καλύτερα. Κύριε Παπα-Νικολάου, συζητούμε την έκθεση για την ε, διαχείριση της επιστροφής, το θέμα το οποίο εσείς εισηγήσετε. Έλεγα λοιπόν ότι ευχαριστώ τον κύριο Νικολάου για την εισηγησή του. Δεν συμφωνούμε πάντοτε αλλά έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε και εδώ και αλλού, σε άλλες επιτροπές. Οπότε μπορούμε να βρούμε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Δεν κατάλαβα πλήρως γιατί το έλεγε ζήτησε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Γιατί δεν περίμενε η Επιτροπή να προβεί σε κάποιο τους απολογισμό για αυτή την οδηγία της επιστροφής και έτσι να διορθωθούν καλύτερα τα πράγματα, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή με τέλος του χρόνου θα είχε συλλέξει πολλά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε πως έχει η κατάσταση και ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα και ότι ακόμα και τα κάποια λίγα θετικά που υπάρχουν από αυτή την ε, οδηγία της ντροπή δεν εφαρμόζονται από όλα τα κρατημέλη. Αυτό έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Επίσης, έχουμε την τύχη σε εισαγωγικά ο ΙΕ να έχει ασχοληθεί με το θέμα. Έχουμε την έκθεση του ειδικού εισηγητή για τα φερμανά δικαιώματα που ασχολείται εκτεταμένα για αυτή την ε, οδηγία της επιστροφής και για τις ε, ε συνέπειες της. Πρόκειται για βασική μέρημα του ΟΗΕ, μια που η κράτηση δεν θα πρέπει ποτέ να είναι η μόνη λύση όσον αφορά τους λάθρομετανάστες. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι έχουμε όλο ένα και περισσότερη κράτησή τους. Πρόκειται για κάποιους που είναι σε καταστασία ευάλωτη, πρόκειται για γυναίκες, για ανηλίκους, για συνόδευτους ανηλίκους. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει έτσι να βλέπουμε τα πράγματα. Επίσης άλλο στοιχείο, όταν έχουμε το κείμενο να υποβάλουμε και κάποιες τροπολογίες, μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο προκυβεί από το έργο του ΟΗΕ και των μη κυβερνήτων οργανώσεων, ότι δηλαδή οι, τα κράτη-μέλη, κυρίως αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην βλέπουν τα πράγματα μόνο από την οπτική της ασφάλειας. Γενικά, μόνο οι υπουργοί εσωτερικών ασχολούνται με το θέμα και ξέρουμε όλοι ότι όταν δεν υπάρχει σφαιρική, συνολική αντιμετώπιση, δεν σημειώνεται πρόοδος. Και το κιασάκι στην τούρτα είναι να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα αριθμητικά στοιχεία. Να μην λέμε ότι πλημμυρίσαμε από μετανάστες. Είδαμε πως η εξέλιξη υπήρξε. 2,5 με 3% τελευταίους έτσι αν είχαμε δώσει την ίδια σημασία στην διακίνηση προσώπων όσο στη διακίνηση εμπορευμάτων, τότε θα ήμασταν σε καλύτερη θέση όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο κύριος Ιακολίνο, για δύο λεπτά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, ιδίως αυτή τη στιγμή. Πολύ καλά το περιέγραψε ο Γιώργος Παπανικολάου και θα πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ των προσφύγων που έχουν δικαίωμα ασύλου, διότι είναι ένα κοινό καθεστώς το οποίο προβλέπεται και με κανόνες τους οποίους εμείς πρόσφατα ως Κοινοβούλιο εγκρίναμε, από τους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι φτάνουν στην Ευρώπη αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παραμένουν στη χώρα. Για τους οικονομικούς μετανάστες υπάρχει υποχρέωση του επαναπατρισμού. Και θα θέλαμε να είναι εθελούσιος αυτός ο επαναπατρισμός για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε καλύτερο εσωτερικό συντονισμό και να υπάρχει μια λογική μεταξύ των διαφόρων ε, υπηρεσιών. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εξωτερική δράση, την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Χρειαζόμαστε συνεργασία με τρίτες χώρε. Αλλά αυτή τη στιγμή που εξακολουθούμε να βιώνουμε αυτές τις τραγωδίες στη Μεσόγειο, πρέπει να ε, διαρθρώσουμε λίγο καλύτερα την υποδοχή. Υπάρχει μια επιστροφή διότι αρχικά τους υποδεχθήκαμε. Οι προσπάθειες λοιπόν που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των ροών, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτούς τους εμπόρους του θανάτου, που πολύ συχνά τροφοδοτούν με χρήματα μια ελπίδα την οποία στη συνέχεια τους την αρνούμαστε εμείς αποφασιστικά, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συνολική διαχείριση. Για τις επιστροφές λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η έκθεση η οποία Ε, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανικολάου. Περιμένουμε την έκθεση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένουμε τουλάχιστον μια ρανίδα ενδιαφέροντος από το Συμβούλιο, διότι πρέπει να νικήσουμε αυτή τη μάχη ε, εναντίον όλων αυτών των ε, λάθρεμπόρων και να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό καταμερισμό του βάρους μεταξύ όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Φλότρ. Για δύο λεπτά. Εγώ νομίζω ότι η προσέγγιση που μπορούμε να επιλέξουμε για να είναι χρήσιμη η δουλειά είναι να εξετάσουμε τα βασικά εργαλεία επιστροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αξιολογήσουμε την εφαρμογή τους από την σκοπιά κυρίως του σεβασμού των ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων βεβαίως και της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν είτε για να κάνουμε προτάσεις νομοθετικές τροποποίησεις είτε να ζητήσουμε την σωστή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων προστασίας των ατόμων που εμπίπτουν στις διαδικασίες αυτές. Υπάρχει και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν οι συμφωνίες της επιστροφής, όπου μπορεί κανείς νομίζω να εξετάσει μόνο τις κοινοτικές και να βασιστεί Εγώ νομίζω ότι ήταν εξαιρετική αξιολόγηση και πολύ επικριτική της ε, Κομισιόν με πολλές ιδιαίτερα χρήσιμες συστάσεις οι οποίες έμειναν όμως σε κάποιο σιρτάρι και τελικά δεν εφαρμόστηκαν. Τουλάχιστον για τις συμφωνίες λοιπόν επιστροφής. Υπάρχει μια εργασία αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να βασιστούμε στην εργασία αυτή για να επανέλθουμε με συστάσεις ή στις συστάσεις εκείνες ή να υποβάλουμε νέες. Ιδίω την δυνατότητα αναστολής των συμφωνιών ή και μάλιστα καταγγελίας τους όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων που εμπίπτουν στο απαιδείο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών να συνεργαστούμε με τους μη κρατικού οργανισμούς των χωρών μελών και στην Μικτή Επιτροπή Επιστροφών που βρίσκεται στην βάση των συμφωνιών αυτών και να έχουμε και την δυνατότητα να παρακολουθούμε την εφαρμογή των διατάξεων προστασίας των ε, ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αν λοιπόν η Κομισιόν διαθέτει νέες πληροφορίες για τις ειδικέ ε, συμφωνίες, για παράδειγμα με το Πακιστάν, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μας τις υποβάλει για να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερο, Frontex. Frontex στην εντολή του μπορεί να επιτρέπει η εντολή του να καλείται να οργανώνει τις επιστροφές, τις συζητήσεις που κάναμε δεν καταφέραμε να επιτύχουμε να γίνεται ξεχωριστό ανεξάρτητο monitoring των δραστηριοτήτων της Frontex. Ωστόσο, έχουμε επιτύχει να φτιαχτεί εντεταλμένος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γραφείο παρακολούθησης ε, της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων που θα μπορούν να οργανώνονται από την ίδια τη Frontex και να λειτουργήσουν τα όργανα αυτά έτσι ώστε να γίνεται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, ο πυρήνας που είναι η ίδια η οδηγία επιστροφής, νομίζω όλοι εδώ έχουμε επισκεφτεί κέντρα κράτησης και έχουμε διαπιστώσει ορισμένες καταστάσεις πραγματικά απερίγραπτες. Κράτηση μάλιστα και κοινοτικών υπηκών που είναι κάτι το σύνηθες ε, τρομερές συνθήκες προσωπικής υγιεινής ανθρώπων που αποστέλλονται πάλι στις πατρίδες τους ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα να, να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα ενώ η κράτηση θα πρέπει να είναι το ίστατο μέτρο και μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερη έχοντας πλέον εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές κάτι που νομίζω ότι πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Επίσης το θέμα της κράτησης των ανηλίκων σε κέντρα κράτησης καθώς επίσης πρόσβαση μη κρατικών οργανισμών και δημοσιογράφων. Έχουμε ήδη υποβάλει σχετική ερώτηση στην Κομισιόν με απάντηση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις εργασίες μας. Νομίζω λοιπόν ότι το σύνολο των ε, θεμάτων αυτών για την αξιολόγηση της σωστής εφαρμογής κυρία Βεζιά ε, Φλότ, Φλότ, κυρία Φλότ, σας παρακαλώ ολοκληρώστε πιο γρήγορα θα τελειώσω αν με αφήσετε. Μου φαίνονται λοιπόν πολύ σωστά για να στήσουμε την αρχιτεκτονική της εργασίας μας. Νομίζω τώρα είναι σημαντικό να ακούσουμε, το, να, να ακούσουμε την Κομισιόν. Και λέγομαι φλότρο στο κάτω της γραφής φτάνουμε πια και στο τέλος της θητείας. Πήρατε πέντε λεφτά. Σας έχω πει, με συγχωρείτε, ζήτησα συγγνώμη για το λάθος το όνομα. Είμαστε ήδη πολύ καστερημένοι και έχω ψηφοφορία. Είναι πολύ απλό να αφήνετε τον λόγο στον εισηγητή και στους σκιώδεις των ε, επιτροπών. Είναι επίσης πολύ απλό. Των ομάδων, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Υπάρχει πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Αλλά χρειάζεται και πολιτική επιστροφής. Και νομίζω ότι είναι καλό πού πάει να γίνει αυτή η προσπάθεια. Ε, ένας αριθμός συναδέλφων πήγαμε σε αποστολή το προηγούμενο καλοκαίρι στην Ισπανία για να εξετάσουμε τις δραστηριότητες της Frontex και τις υπηρεσίες της ακτοφυλακής. Μας είπαν ότι στους 10 που έρχονται στην Ισπανία από την Μεσόγειο, ένας μόνο θα κρυθεί ε, ότι ζητεί άσυλο, ένας θα επιστραφεί και οι υπόλοιποι 8 εξαφανίζονται στη χώρα. Αυτό συμβαίνει με αυτούς που καταφθάνουν παράνομα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επιστρέφονται. Θεωρώ ότι θέτει ένα μέγα πρόβλημα για την πολιτική αυτή και για την εργασία μας. Πρέπει να φτιάξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία σαμποτάρεται ωστόσο και από μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά υπάρχει και μια αντίσταση των κυβερνήσεων και των αριστερών κομμάτων που βρίσκουν όλο και περισσότερες δικαιολογίες για να μην στέλνουν τους ανθρώπους αυτούς πίσω στις χώρες προέλευσής τους και από την άλλη μεριά υπάρχει πολύ περιορισμένη συνεργασία και μάλιστα και μια ενεργός αντίσταση από την πλευρά των χωρών εκείνων από όπου προέρχονται οι μετανάστες αυτοί. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να επιβληθούν κυρώσεις, να προβλέπονται κυρώσεις. βέβαια υπάρχουν οι συμφωνίες επιστροφής με τρίτες χώρες. Αλλά οι χώρες οι οποίες δεν σέβονται τις υποχρώσεις τους πρέπει να υποστούν κυρώσεις. Για παράδειγμα, σκέφτομαι τις πιστώσεις στην πολιτική της γειτονίας. Θα πρέπει να παγώσουν οι πιστώσεις αυτές όταν διαπιστώσουμε ότι μια τρίτη χώρα δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει μέσω, της, ε, μέσω των συμφωνιών επιστροφής. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή θα πρέπει, εφόσον δεν λειτουργούν οι ενωσιακές συμφωνίες, να περάσουμε σε διμερείς συμφωνίες. Τώρα η Κομισιόν και το Συμβούλιο να απαντήσετε στον ε, εισηγητή, αλλά πάρα πολύ σύντομα. Έχετε το λόγο να Έχετε το δικαίωμα να τοποθετηθείτε, αλλά πραγματικά συντομότατα η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η Κομισιόν κατά πάσα πιθανότητα στις 17 Δεκεμβρίου θα υποβάλει την πρώτη της έκθεση εφαρμογής για την ε, οδηγία ε, επιστροφής. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι η έκθεση αυτή θα έχει θετικό χαρακτήρα, θα δηλώνει ότι στην πράξη η Συμφωνία Επιστροφής έχει συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή που καλύπτει. Πιο συγκεκριμένα θα αναλύουμε στην έκθεση αυτή τα περισσότερα από τα θέματα που ανέφεραν τα αξιότιμα μέλη στις παρεμβάσεις τους. Θα μιλούμε δηλαδή για κράτηση, για εναλλακτικές επιλογές στην κράτηση, για την παρακολούθηση, το monitoring δηλαδή των αναγκαστικών επιστροφών της ε, επιχειρήσης Frontex, την αποτελεσματικότητα την ε, ποινικοποίηση και ούτω καθεξής. Αυτά όλα τα θέματα θα τα θέσουμε και θα κάνουμε και ορισμένες συστάσεις πολιτικής. Εν ώψη αυτού του ιστορικού προβληματιζόμαστε λίγο που βλέπουμε ότι η έκθεση αυτή πρωτοβουλία πάει να κάνει το ίδιο πράγμα και ταυτόχρονα. Αυτή είναι η πιο μεγάλη μας ανησυχία. Κατά τη γνώμη μας θα ήταν καλύτερα να περιμένετε μέχρι ότου μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε την έκθεσή μας περί εφαρμογής και εκεί τότε να υπάρξει μια σταθερή βάση, μια στέρεα βάση για να ε, συζητήσετε. Το Συμβούλιο. Όχι, δεν απαραίτητο. Καλά, ευχαριστώ. Κύριε Σεγητά, σύντομα. Very shortly, ε, Σύντομα κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις και επίσης να απαντήσω στην κυρία Βερζιά. Η αρχική προσέγγιση και το πνεύμα που διαπνεί την προσέγγιση μέσα να έχουμε τη συνολική εικόνα και να αναρωτηθούμε κατά πόσον μπορούμε να έχουμε μια τέτοια συνολική προσέγγιση όσον αφορά την διαχείριση των επιστροφών. Μια πτυχή αυτού του θέματος είναι η υλοποίηση, εφαρμογή της οδηγίας για τις επιστροφές. Έχουμε την πρόταση επίσης και από τις άλλες πολιτικές ομάδες να καλυφθεί και αυτή η οδηγία και γι' αυτό και την εντάξαμε εδώ. Σκοπός μας δεν ήταν να προσπαθήσουμε και να δουλέψουμε παράλληλα και κατ' επικάλυψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι να καταλήξουμε στο να πριν τα ανέβει η σύγχυση. Αυτό σας να κάνουμε, να αναρωτηθούμε αν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια συνολική προσέγγιση ό,τι συμφωνείτε να εφαρμόζετε και να τηρείτε. Να έχουμε όλα τα μέσα που χρειάζονται, ούτω ώστε να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση της επιστροφής. Δεν το έχουμε αυτό. Αλλά θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αποκτήσει κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, όλους τους κοιόδες για τη συνεργασία τους. Πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε προτεραιότητες, να μπορούμε σε κάποια συνάντηση να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στα πιο βασικά για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την ε, παραβίασή του, όποτε έχουμε τέτοιε περιπτώσει που δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Γιατί έχουμε και κάποια παράκαμψη των συμφωνιών, έχουμε διάφορα τέτοια ζητήματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Οπότε σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Οπότε παρακαλώ πρόεδρε να μπορέσουμε το σύντομο δυνατόν να προχωρήσουμε και να σας ε, παρουσιάσουμε το σχέδιο της έκθεσης. Τώρα, έχουμε αυτές τις τελικές σκέψεις του εισηγητή. 27 δεκάτου θα παρουσιαστεί και, και προθεσμία είναι 5 δεκάτου για τις τροπολογίες και 22 Ιανουαρίου η ψηφοφορία. Συμφωνείτε. Πάμε στις ψηφοφορίες τώρα. Τρεις ψηφοφορίες έχουμε και έχουμε καθυστερήσει. Δεν είναι δύσκολα, αλλά είναι τρία. Τρία θέματα. Έχετε διαδικαστικό. Κύριο Ζέλστρο. Υπάρχει κάποια προβλήματα με τις λίστες για την ψηφορία. Αφήστε που εγώ δεν πήρα καν έγκαιρα την λίστα για την ψηφορία. Ψάχνω, τις τελευταίες μέρες τίποτα δεν έγινε. Έχω μάλιστα γράψει και κάποιο γράμμα σχετικά. Και από ό,τι ξέρουμε πρέπει να αναβάλει ψηφορία αν δεν έχουν λίστα ψηφορίας τα μέλη. Νομίζω ότι κάθε ψήφος έχει σημασία. Και μου υποσχέθηκαν ότι θα μου έχουν δώσει αυτόν τον κατάλογο έγκαιρα. Τι να σας πω. Οι υποσχέσεις που δίνονται στις Βρυξέλλες δεν τηρούνται. Πρόεδρος. Έτσι γίνεται. Συνήθως. Δεν έχω ακούσει τέτοιου είδους παράπονα. Όλοι στην Λίμπε λαμβάνει τον κατάλογο τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Και χθε αυτό έγινε. 24 ώρες πριν λάβατε όλοι τον κατάλογο. Και θα λέμε πως αυτό το οποίο είπατε, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτε παράπονα. Όχι, εγώ έχω παραπονεθεί, Πρόεδρε, τακτικά για το θέμα αυτό. Και πολλές φορές το έχω πάρει μισή ώρα πριν την ε, συνεδρίαση. Είναι τρομερό. Όλοι οι υπόλοιποι έλαβαν τους καταλόγους χωρίς πρόβλημα. Πάντως θα λεφθεί υπόψη αυτό το οποίο είπατε. Πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Και να διεξαγάμε τις εφορίες. Εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων. Έλεγχος κρατών μελών. Άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων επιτροπής. Μπένοβα είναι η Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έχουμε στην πρώτη παράγραφο μια τεχνική διόρθωση. Πίνει υπέρ, πίνει κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Δεν Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, λέει ο Πρόεδρος. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Δεν έχετε κάρτα. Τότε θα ψηφίσουμε. Τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία ε, ναι, 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αιτιολογική παράγραφος Γ τροπολογία 3. Ναι, ναι, τροπολογία 2. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 38 ψηφί υπέρ, συνεδρίες κυρία Μπένοβα και τώρα ε, το, το σχέδιο του πρωτοκόλου για, την, για τις παράνομη κατασκευή και διακίνηση πυροβολών όπλων. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ματιέ. Σχεδόν χωρίς τροπολογίες. Επομένως ψηφίζουμε το τελικό κείμενο. Ψηφίζουμε. Με ηλεκτρονικό τρόπο. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. 40. Μία ε, αποχή, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια κυρία Ματιέ. Και τώρα η τρίτη ψηφοφορία. Αφορά την έκθεση του συναδέλφου Κλάς. Που αφορά την τροποποίηση τη απόφαση σε σχέση με κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τα οποία βγήκε η Ευρωπόλ στην αυτή συμφωνία. Ψηφίζουμε τι τροπολογίε. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ε, αποσύρεται, καταπίπτει, αποσύρεται, άρα πάμε στην τελική ψηφοφορία του κειμένου. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Σαράντα υπέρ. Χωρί αποχέ, ποιου κατά, συγχαρητήρια κύριε Κλάς. Πάμε παρακάτω μετά την ψηφοφορία. Σημείο 10. Είναι έλεγχος προσώπων στα εξωτερικά σύνορα. Μονομερής αναγνώριση Κροατίας και Κύπρου ισοδυνάμων εγγράφων. Ισοδυνάμων με τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Για πρόθεση διαμονής στην επικράτεια μέχρι 90 μέρες σε με 180 μερών. Τάνια Φαζόν είναι η συγκίτρια. Δεν παρίσταται. Κύριε Μωράξη, μπορεί να λέτε το λόγο για λογαριασμό της εισηγητρίας και κατόπιν θα ακούσουμε τους βουλευτές στην Επιτροπή και την Προεδρία. Πρώτα από τον κύριο Μωράης όμως, λογαριασμό της κυρίας Φαγιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Φαζόν δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα λάβει πρώτα το λόγο η Επιτροπή. Να ξεκινήσω. Ναι, μισό λεπτό. Βάσει τη διαδικασία θα πρέπει πρώτα να λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα μιλήσει ο κύριο Μωράη εκ μέρου τη εισηγήτρια τη κυρία Φατζάν και μετά οι σκιώδει και τα υπόλοιπα μέλη. Αν θέλει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο να μα παρουσιάσει το θέμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που διαβάσετε ήδη τον πολύ μακροσκελή και περίπλοκο τίτλο αυτού του θέματος το οποίο κλήθηκα να σας παρουσιάσω σήμερα. Καταρχάς να σας εξηγήσω λίγο το γενικό πλαίσιο της πρότασης και γιατί υποβάλλει σχετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να το αναλύσουμε αυτό και κατόπιν να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία-τέσσερα θέματα πιο συγκεκριμένα. Να ξεκινήσω με το γενικό πλαίσιο να υπενθυμίσω ότι όταν ένα νέο κράτος μέλος εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται αυτομάτως ε, μέλος της ε, Σέγγεν. Συνήθως ε, περνά ένα χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνία προσχώρησης ενός κράτους μέλους και της άρσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα μεταξύ του χώρου Σέγγεν και του νέου κράτους μέλους συνθήκες προσχώρησης προσφέρουν μια διτή διαδικασία του κεκτημένου Σέγγεν για τα νέα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποια τμήματα του κεκτημένου Σέγγεν τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν από την ημέρα της προσχώρησης. Κάποια άλλα τμήματα του κεκτημένου Σέγγεν εφαρμόζονται μόνο την ημερομηνία που το κράτος μέλος εντάσσεται στο χώρο Σέγγεν. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι στον τομέα των θεωρήσεων διαβατηρίων υπάρχει περιορισμένος αριθμός μέσων του κεκτημένου Σέγγεν που εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία και πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησής τους. Και να επιστήσω κυρίως την προσοχή σας στον κανονισμό 539 του 2001, τον οποίο έχετε επίσης προς τροποποίηση ε, στα έγγραφά σας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει υποχρέωση θεώρησης για όλες ε, τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στον αρνητικό κατάλογο, δηλαδή της έλλειψης υποχρέωσης θεώρησης ε, από την ημέρα προσχώρησης. Υπάρχουν κάποιες άλλες διατάξεις οι οποίες δεν ισχύουν από την ημέρα προσχώρησης. Βάσει του κώδικα θεωρήσεων, ένα κράτος μέλος δεν συνδέεται αυτόματα με το σύστημα VIS, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις του κεκτημένου Σέγγεν για την αμοιβαία αναγνώριση των θεωρήσεων. Αφενός λοιπόν στην περίπτωσή μας η Κροατία πρέπει να επιβάλλει ε, υποχρέωση θεωρήσεων διαβατηρίων για τις χώρες οι οποίες ε, πρέπει να έχουν θεώρηση διαβατηρίων βάσει του κανονισμού 539 του 2001, αλλά η αμοιβαία αναγνώριση δεν ισχύει ακόμα. Και αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωσή μας η Κροατία θα πρέπει να ζητά θεώρηση διαβατηρίου, ακόμα και αν αυτός ο οποίος θέλει να ταξιδέψει στην ε, Κροατία διαθέτει μία θεώρηση πολλαπλών εισόδων για τις υπόλοιπες χώρες Σέγγεν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αύξηση ε, στο φόρτο εργασίας, ο οποίο δεν είναι αιτιολογημένος. Διότι κάποιο ο οποίο έχει θεώρηση Σέγγεν ή έχει μια άδεια παραμονής ε, σε χώρα Σέγγεν, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αποτελούν ε, ύποπτους παράνομη μετανάστευση σε νέα κράτη-μέλη όπω είναι η Κροατία. Για το λόγο αυτό λοιπόν, ώστε να μην έχουμε περί τη γραφειοκρατία, ήδη από το παρελθόν για τις χώρες οι οποίες εντάχθηκαν το 2004 και το 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κάποια μέσα τα οποία επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν μονομερώς τις θεωρήσεις διαβατηρίων χώρου Σέγγεν και τις ε, άδειες παραμονής ε, για ε, ένα διάστημα στη χώρα τους. Αυτή η διάταξη εδώ θέλει να προσφέρει την ίδια δυνατότητα στην Κροατία. Να μπορεί η Κροατία δηλαδή να αναγνωρίσει μονομερώς ε, τις θεωρήσεις ε, διαβατηρίων Σέγγεν και τις άδειες παραμονής Σέγγεν. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, το σκεπτικό μας είναι ότι και για το Συμβούλιο και για τα κράτη-μέλη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα ε, για λόγους αρχής. πρόκειται απλώς για επανάληψη μιας διαδικασίας η οποία έχει γίνει άλλε δύο φορέ στο παρελθόν. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τώρα, κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ε, αντίστοιχες αποφάσεις. Οι αποφάσεις εκείνες ε, επέτρεπαν μονομορή αναγνώριση θεωρήσεων διαβατηρίων και ε, διαμονής μόνο για διέλευση μέσω του νέου κράτους μέλους. Εάν κάποιος υπήκος τρίτης χώρα ήθελε να πάει στο νέο κράτο μέλος για να κάνει ένα μήνα διακοπές, τότε δεν ίσχυε η μονομορή αναγνώριση, διότι θεωρείται ότι σε αυτή την περίπτωση το νέο κράτο μέλος είναι ο βασικός προορισμό του ταξιδιού και επομένως θα πρέπει ε, να υπάρχει διαδικασία θεώρησης και να υποβάλλεται αίτηση και επεξεργασία. Ο κώδικας των θεωρήσεων ε, δεν έχει πλέον ε, θεώρηση διέλευσης. Υπάρχει μία θεώρηση Σέγγεν που χρησιμοποιείται είτε για διέλευση είτε για σύντομη διαμονή. Ακριβώς βάσει αυτής της λογικός λοιπόν η πρόταση επιτρέπει στην Κροατία να αναγνωρίσει μονομερώς θεωρήσεις διαβατηρίων και άδειες διαμονής για μικρό διάστημα στην επικράτειά τους. Κάποιο λοιπόν ο οποίος έχει θεώρηση διαβατηρίου πολλαπλών εισόδων μπορεί να πάει στην Κροατία αν η Κροατία αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα χωρίς να απαιτείται να αποκτήσει μια θεώρηση ε, για ε, μικρό διάστημα ε, σύντομης ε, διαμονής της Κροατίας. Πρόκειται λοιπόν για μια μικρή αλλαγή που έχει προκύψει από τον κώδικα θεωρήσεων και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να ανακαλέσουμε τις προηγούμενες αποφάσεις οι οποίες ισχύουν ακόμα για την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για να υπάρχει επέκταση της δυνατότητας να αναγνωρίζονται μονομερώς οι θεωρήσεις όχι μόνο για διέλευση αλλά και για σύντομη διαμονή. Μια τρίτη παρατήρηση γιατί αναφέρουμε στον τίτλο μόνο την Κύπρο και την Κροατία και όχι και τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Διότι προς το παρόν δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στη Σέγγεν. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση, Είχαμε θεωρήσει ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν σύντομα και επομένω ε, θα ήταν λανθασμένο πολιτικό μήνυμα στην πρόταση αυτή να καλύπτονται ακόμα και η Ρουμανία και η Βουλγαρία διότι για αυτέ, αυτή τη στιγμή θα ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν ισχύουν οι συνήθει κανόνε ε, Σέγγεν για την αναγνώριση των θεωρήσεων διαβατηρίων και ούτω καθεξής. Δεν θέλαμε να δώσουμε λοιπόν την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όταν θα εγκριθεί η πρόταση η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν θα είναι ακόμα στο χώρο Σέγγεν. Βεβαίως, όταν θα φτάσουμε στη στιγμή της έγκρισης της πρότασης, εάν μέχρι τότε η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν, τότε θα πρέπει να τις προσθέσουμε στην πρόταση. Που σημαίνει, αν απλουστεύσω λίγο τα πράγματα, εκεί που λέει τώρα Κροατία και Κύπρος, ε, μπορούν να αναγνωρίσουν μονομερούς, θα έχουμε Κροατία, Κύπρος, Ρουμανία και Βουλγαρία. Μια τεχνική προσαρμογή λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Μια τελευταία παρατήρηση για το κοσμοπέδιο. Συνήθως δίνεται έγκριση στο νέο κράτος μέλος να αναγνωρίζει έγγραφα τα οποία επιτρέπουν ε, σε κάποιον να ταξιδεύει σε όλο το χώρο Σέγγεν. Ε, θεωρήσεις διαβατηρίων ή άδειες διαμονής οι οποίες εκδίδονται από χώρα Σέγγεν. Να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι οι Κωσοβάροι πολίτες Καταρχήν, δεν θα έπρεπε να έχουν θεώρηση η οποία να ισχύει για όλο το χώρο Σέγγεν. Όπω γνωρίζετε, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν αναγνωρίζουν το κοσμοπέδιο και επομένω αυτό έχει συνέπειε και για τη θεώρηση η οποία εκδίδεται. Αν είναι κράτο μέλο το οποίο δεν αναγνωρίζει το κοσμοπέδιο, θα εκδώσει θεώρηση ε, θεωρήσεις οι οποίες αποκαλούνται LTV, περιορισμένης ε, γεωγραφική ε, επικράτειας δηλαδή, διότι επιτρέπεται να ταξιδέψουν μόνο συγκεκριμένες περιοχές. Εάν εκδίδεται θεώρηση από χώρα που αναγνωρίζει το κοσυφοπαίδιο και οι περισσότερες χώρες το αναγνωρίζουν, τότε θα είναι θεώρηση Σέγγεν που θα επιτρέπει σε κάποιον να ταξιδεύει σε όλο το χώρο Σέγγεν, εκτός τη επικράτεια των χωρών που δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπαίδιο. Επομένω, η θεώρηση αυτή έχει ε, συγκεκριμένη εδαφική ε, ισχύει και δεν καλύπτει όλο το χώρο Σέγγεν. Για να μην αποκλειστεί λοιπόν ε, ε, και το Κωσυφοπέδιο από αυτή τη δυνατότητα και οι Κωσοβάροι πολίτες, ε, προβλέπεται στο κείμενο και θα το βρείτε αυτό και στις προηγούμενες αποφάσεις, διότι ε, μάλλον δεν θα το βρείτε γιατί το θέμα του Κωσυφοπεδίου δεν είχε προκύψει ακόμα, ε, επιτρέπεται λοιπόν μονομερής αναγνώριση έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων σε κοσοβάρους πολίτες η οποία ισχύει για όλο το χώρο Σέγγεν με την εξαίρεση των χωρών που δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπαίδιο. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση. Επειδή υπάρχουν αντίστοιχε αποφάσει οι οποίε έχουν εγκριθεί στο παρελθόν, φαντάζομαι ότι δεν θα ε, υπάρξουν προβλήματα με τη συγκεκριμένη πρόταση. Ωραία. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Μωράε, εκ μέρου τη κυρία Φαγιών που είναι η συγγήτρια. Κλοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Φαζόν δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Συζήτησα το θέμα αυτό μαζί της και η προσέγγιση της είναι απλή. Όσον αφορά την ουσία, θεωρεί ότι μετά από την προσχώρηση των χωρών το 2004 και το 2007 το θέμα αυτό είναι τεχνικής φύσεως, αρκετά απλό και νομίζω ότι η ομάδα θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετώπισαν μια πολύ περίπλοκη κατάσταση με τον κανονισμό 539 του 2001 που αναφέρθηκε στην παρουσίαση του εκπροσώπου της Επιτροπής. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα εδώ για ένα τόσο τεχνικό ζήτημα. Αυτή είναι κατά βάση προσέγγισή μας. Τώρα η συζήτηση μπορεί να διευρυνθεί για την ε, Ρουμανία και τη Βουλγαρία που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην, ε, ε, στο χώρο Σέγγεν και ίσως μπορεί να διευρυνθεί η συζήτηση λόγω αυτού και να θέλουν οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία αλλά για την Κροατία είναι μάλλον απλά τα πράγματα, δεν θα πρέπει να υπάρξουν προβλήματα το απλουστευμένο καθεστώς το οποίο καθορίστηκε το 2004-2007 για την προσχώρηση των νέων χωρών είναι το αντίστοιχο καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται εδώ. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα, θεωρούμε ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα και μια τεχνική προσέγγιση. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιπλοκές και αυτή είναι και η προσέγγιση της κυρίας Φαζόν. Επειδή όμως υπάρχει το θέμα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο για τα θέματα αυτά. Νομίζω όμως ότι για μα και για την κυρία Φαζόν είναι απλό το θέμα και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή του και τη δουλειά του για το θέμα αυτό μέχρι τούδε. Ωραία. Τα μέλη τώρα. Ο κύριος Πλάνκοβιτς. Παρακαλώ. θέλει το χέρι του Κύριε Ντανάκα, βλέπω. Κύριε Πλάκοβιτ, έχετε πρώτα στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω επίση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι επεξηγήσει όσον αφορά τι προτάσει τη για αυτή την σημαντική απόφαση που πραγματικά θα πλουστεύσει τι διαδικασίε για την Κροατία ω νέο κράτο μέλο για την μονομερή αναγνώριση αυτών των θεωρήσεων διαβατηρίων όσον αφορά την ε, σύντομη διαμονή επίση και τι ε, βίζε διαμετακόβηση που είναι πάρα πολύ χρήσιμο να καταργήσουμε κάποιο είδους ε, περιττές γραφειοκρατίες για κάποιους θαγενείς τέτοιων χώρων. Πρώτα απ' όσον αφορά τον στρατηγικό μα στόχο μετά την ε, ε, προσχώρηση και επίσης για την προοπτική του να μπούμε στο Σανγκέν και να μπορούμε να πληρούμε τα αναγκαία κριτήρια διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μια χώρα η οποία έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική των διορίσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο συντομότερο είμαστε μέλος του χώρου τόσο καλύτερα. Γιατί είμαστε σε μια μεσοβέζικη κατάσταση. Ε, μισό μέσα, μισό έξω και βέβαια είναι, έχει σημασία αυτό γιατί έχουμε πολύ τουρισμό και έχουμε διάφορους που έρχονται και από Τουρκία. Τέλος πάντων όλα αυτά, ιδίω το καλοκαίρι θα έχουν σημασία. και ο κόσμος περιμένει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί όπως θα θυμάστε είχαμε συμφωνήσει πρώτα πρώτα την, την δόση των 40 ε, εκατομμύρια το 2013 και επίσης είπαμε για 2014 θα έχουμε 80 εκατομμύρια που επρίχνουμε και αυτά τα χρήματα να τα βάλουμε, να τα λάβουμε ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει τα λάθη όπως εκείνο το λάθος όσον αφορά τον περιορισμό ε, όσον αφορά αυτό το οποίο έγινε με την παραγραφή του του σύλληψη, Τέλο πάντων, αυτό το οποίο χρειάζεται Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι όλα αυτά εν ευθέτω χρόνο θα εγκριθούν και θα διευθετηθούν. Και σα ευχαριστούμε την εισήγησή σα. Είναι θα περιμένετε να λάβετε το λόγο μετά τους ε, σιώδες. Ναι, ναι, ναι, να λάβω το λόγο, γιατί ε, είναι τεχνοκρατικό, τεχνικό το ζήτημα και ευχαριστούμε πάρα πολύ το, τον εισηγητή που μας τα εξήγησε τόσο πολύ, γιατί μια που είναι τεχνικό το θέμα, είναι πάρα πολύ βασικό ε, ο κόσμος να μπορέσει να το καταλάβει βοηθάει πάρα πολύ το θέμα του, το, το, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η οποία θέλει να μπει στο Σέγγεν. Και βέβαια το ίδιο ισχύει ε, σαν θετικό αποτέλεσμα και για την Κροατία. Is that how you pronounce it, Σβίκα? Σβίκα, Σφίκα. Είναι το όνομά σας, ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Από πλευρά της κροατικής συνιστώσης συνιστώ, ε, συμφωνώ συγγνώμη, με όσα όλα λέγθησαν και να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια προς το παρόν. Ζητούμε θεωρήσεις διαβατήριων, αλλά δεν ισχύει η αρχή της αμοιβαίας ε, αναγνώριση. Ε, νομίζω ότι τώρα θα έχουμε λιγότερο, λιγότερο βάρος, λιγότερη δουλειά, Και άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα επιλύσουμε αυτό το ζήτημα σε σχέση με τα όσα θα ζητεί το Σέγγεν. <clears throat> Τώρα τέλος πάντων θα απαλλαγούμε κάποιες αχρήσεις διαδικασίες ο κ. Πλάνκοβιτς και τελικά ο απότερος στόχος της κροατία είναι βέβαια να μπει στο χώρο Σέγγεν. Επομένως η διευκολύνση του Σέγγεν όπως θέλουμε θα ισχύσουν σύντομα. Αλλά βέβαια απόκειται και στην κυβέρνησή μας να εφαρμόσει ε, τις διευκολύνσεις Σέγγεν το Οπότε δεν μπορούμε να παραφερήσουμε θετική αυτή την μονομερή αναγνώριση των θεωρήσεων διαβατήριων. Αφορά μόνο μικρή περίοδο διαμονής, ε, αφορά ε, διαμετακόμιση, αφορά διάστημα 180 ημερών. Δεν είχε κάτι μέχρι σήμερα. Άρα θέλουμε θετική αυτή την πρόταση. Να ισχύσει αυτό το μέτρο χωρίς χωριστή θεώρηση διαβατηρίου. Άλλη. Επίσης σας τονίζω ότι η διαδικασία έχει αρνητικό χαρακτήρα, έχει αρνητικέ επιπτώσει στον τουρισμό. Ο τουρισμός μας πέρσι επλήγει σοβαρά, σημαντικά. Τουρκία, από Τουρκία, από Ρωσία. Ε, ήρθαν λιγότεροι τουρίστες. Οπότε, χαιρετίζουμε την πρόταση. Και θα την επιψηφίσουμε και εδώ και στην Ολομέλη. Μετά από εσάς, θέλει άλλο συνάδελφος να σχολιάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δάλλος. Κύριε Μωράης, εσείς εκ μέρους της κυρίας Φαγιών. Οπότε 27 και 28 Νοεμβρίου θα παρουσιάσουμε την ε, έκθεση και 18-12 προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Συμφωνείτε? Ωραία. Πάμε τώρα στο 11. επιτήρηση εξωτερικών θαλασσίων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρηματική συνεργασίας. Frontex έχει αναλάβει τον συντονισμό στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών. ο οποίος θα αναπτύξει το σχέδιο εκθέσεώς του. Βεβαίως ακόμα πιο σημαντικό τώρα που έχουμε ε, υπόψη μας τα τελευταία τραγικά συμβάντα έξω από το νησί Λαμπεντούσα καθώς και τις ε, έκτακτες αυτές ε, επιχειρήσεις διάσωσης που αναπτύσσει τώρα η Ιταλική κυβέρνηση και ζητεί για αυτές συνεργασία και από άλλες χώρες μέλη καθώς και από τα ευρωπαϊκά όργανα. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τι θα πει ο κ. Σκοέριο και μετά να ακούσουμε την Κομισιόν και την Προεδρία. Εσείς κύριε Κοέλιο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρωτίστως ε, μας ενδιαφέρει να διαφυλάξουμε την ζώνη δικαιοσύνης και ελευθερίας. Άρα χρειαζόμαστε κοινή προσέγγιση για το θέμα της προστασίας των συνόρων, αποτελεσματικούς ελέγχους δηλαδή. Αυτό είναι κέριο. Επίσης, πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας των συνόρων, που όμως δεν πρέπει να υπονομεύει την υποχρέωσή μας να προφυλάσσουμε, να προστατεύουμε τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες των ε, προσώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της δηλαδή πρέπει να φροντίζουν για την προστασία αυτή. Εσείς κύριε Πρόεδρε είπατε, αναφερθήκατε στην τραγωδία της Λαμπεντούσα. Τις τελευταίες μέρες εκατοντάδες άνθρωποι χάθηκαν και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις 25% των ανθρώπων που διασχίζουν τη Μεσόγειο ε, μέσα σε αυτά τα ανασφαλή πλοιάρια τελικά ε, πνίγονται στη θάλασσα. Μερικούς, για μερικούς μάλλον ακούμε. Για άλλα θύματα μόνο μπορούμε να μαντεύσουμε. Η διάσωση των ανθρώπινων ζώων ποτέ δεν πρέπει να αμφισβητηθεί. Ανεξαρτήτως ε, του πλοίου που ζητεί την ε, βοήθειά μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιες τροποποιήσεις στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Γνωρίζουμε ότι η ροή μεταναστών έχει σοβαρότητες επιπτώσεις σε ορισμένες νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γνωρίζουμε επίσης ότι το φαινόμενο ε, αυτό επιβαρύνει και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για ευθύνη, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για λυγγί διότι αυτό αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να διαφυλαχθούν τα ε, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των προσώπων που ζητούν άσυλο. Οι προτάσεις της εκθέσεως μου βασίζονται σε τρεις βασικές αρχές. Γι' αυτό και τη χωρίζω σε τρία τμήματα. Θέλουμε πρώτα δεσμευτικά νομικά εργαλεία, δεύτερον προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τρίτο την αρχή της αλληλεγγύης. η έγκριση δεσμευτικού, δεσμευτικών κανόνων είναι πρώτη της, κυριαρχή, πρώτης της ε, στόχου ε, προτεραιότητας. Τους ίδιους στόχους έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και η ε, απόφαση του Συμβουλίου που ανατράπηκε ωστόσο από το δικαστήριο. Πάντως, εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ναυτικών επιχειρήσεων της Frontex, χρειαζόμαστε, όπως είπα, δεσμευτικούς κανόνες. Εκφράζω πάντως τη λύπη μου, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με ορισμένες δηλώσεις χωρών μελών στο Συμβούλιο. Ορισμένες εξ αυτών απορρίπτουν την ιδέα της νομικής δεσμευτικότητας. Ορισμένες χώρες στο Συμβούλιο δήλωσαν ότι δεν είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει άποψη για τα θέματα αυτά, διότι θεωρούν ότι αυτά είναι καθαρά εθνικής κυριαρχίας. Οι ίδιες χώρες μέλη που δημόσια δήλωσαν ότι διαφωνούν με την απόφαση του δικαστηρίου που επιβάλλει την συναπόφαση. Να λοιπόν πάλι άλλη μια φορά όπου σε θέματα Σέγγεν το Συμβούλιο αποδείχνεται διστακτικό να δεχθεί τον συνομοθετικό ρόλο του ε, Κοινοβουλίου. Εγώ εκφράζω τη λύπη μου σαφώς για τις απόψεις αυτές τις οποίες απορρίπτω και θεωρώ αξιόμεντες. Η Προεδρία θέλει να δώσει προτεραιότητα στο αυτό. Και εδώ σημειώνω εγώ μια αντίφαση με τις δηλώσεις των υπουργών που αφενός εκφράζουν τη λύπη τους για τις εξελίξεις αυτές, από την άλλη μεριά ε, δείχνουν μια διστακτικότητα στην ψήφιση νομοθεσίας η οποία εν τέλει θα ε, επιτρέψει την διάσωση ανθρώπινων ζώων. Δεύτερο, στην έκθεσή μου ζητώ να προωθηθεί η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπου το πιο σημαντικό είναι το δικαίωμα της μη επιστροφής. Η αρχή αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και να λησμονείται επειδή βολεύει ορισμένους σε άλλες περιπτώσεις. Τέλος, ενίσχυση της αρχής της ελεγγύης. Γνωρίζουμε ότι την βασική ευθύνη για τη δημιουργία των συστημάτων ασύλου και τη διαχείριση των συνόρων, επαναλαμβάνω η βασική ευθύνη ανήκει στις χώρες μέλη. Όμως, σε μια περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα, δεν ε, ε, χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένα κοινό σύστημα ασύλου και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα ε, διαχείριση των συνόρων. Άρα εδώ χρειάζονται ορισμένε τροποποίησεις. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία που θέλω να θίξω στην ε, έκθεσή μου κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. From the Commission and the Council. Τώρα Κομισιόν και Συμβούλιο. Ε, κύριε Νίλσεν, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια ένα από τα μέτρα τα οποία συζητούνται μετά από τις ανθρωπιστικές τραγωδίες στα νότια σύνορα της Ένωσης που είδαμε πρόσφατα και τις οποίες προωθεί η κυρία Μάνστρομ είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων Frontex στην περιοχή αυτή και η προσφορά ενίσχυση στις χώρες μέλη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές. Για ε, την πρόθεση των επιχειρήσεων αυτών βλέπουμε την έκθεσή σας ως ε, κύριο εργαλείο γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να σώσουμε όσο δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ταχύτητα με την οποία προωθεί το θέμα η Επιτροπή σας και ευχαριστώ τον εισηγητή σας για την ε, υποστήριξη που δίνει στις προσπάθειές μας. Το σχέδιό του δεν ε, απαιτεί ιδιαίτερα σχόλια από εμά. Ελπίζω μόνο το Συμβούλιο να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σινκεβίτσιους, εκπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, αλλά δεν έχει μικρόφωνο ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Ναι, τώρα εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Στις 5 Σεπτεμβρίου ενημερώσαμε την Επιτροπή σας για τη συνεχιζόμενη εργασία για το σημαντικό αυτό θέμα στις αρμόδιες ε, ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Με την παρούσα ευκαιρία θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις, αλλά πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο καθώς και όλη την Επιτροπή σας για την ταχεία επεξεργασία του σχεδίου εκθέσεως. Ταυτόχρονα επιθυμώ να σας βεβαιώσω ότι η Προεδρία επίσης κάνει πάντα το δυνατό για να διασφαλίσει ότι η θέση του Συμβουλίου θα διαμορφωθεί το δυνατόν συντομότερο. Η Λιθουανική Προεδρία έχει ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση της προτάσεως. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα υποβληθούν στην, στην συνεδρία στη Σκύφα την επόμενη εβδομάδα. Η Προεδρία συντάσσει τώρα το αναθεωρημένο κείμενο της ε, προτάσεως και ο δεύτερος γύρος συζητήσεων θα γίνει στην ομάδα εργασίας συνόρων τον Νοέμβριο. Η αποφάσεις που θα λάβουμε μετά για το πώς θα προτείνουμε να συνεχιστεί η εξέταση του σχεδίου, του σχεδίου κανονισμού εννοείται, στις αρμόδιες ε, ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και στο Συμβούλιο, θα εξαρτηθεί από την πορεία αυτών των συζητήσεων. Εάν οι συζητήσεις αυτές αποβούν επιτυχής, θα ζητήσουμε εντολή στην Κορεπέρ 2 για την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως λέχθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου στις 5 Ενάτου, τα πιο ευαίσθητα άρθρα είναι τα 9 και 10. Ορισμένες χώρες μέλη πρότειναν τα άρθρα 9 και 10 της προτάσεως να γίνουν συντομότερα για να αναφέρονται ευθέως στο διεθνές δίκαιο και στο σχέδιο επιχειρήσεως της κάθε επιχειρήσεως. Θα κάνει η Προεδρία μας κάθε τι το δυνατό για να πετύχει συμβιβασμό. Βέβαια, διαβεβαιώνουμε την Επιτροπή σας ότι η Προεδρία θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που δίνει στο σχέδιο εκθέσεώς της η Επιτροπή σας στη διάρκεια της επεξεργασίας της ε, προτάσεώς μας. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μου. Ευχαριστώ. Τώρα έχω ορισμένα μέλη, λέει ο Πρόεδρος. Η λίστα... Κύριος Χέλζερ πρώτος. Σκιώδης πρώτα, Σκιώδης πρώτα. Χόλτσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. βασική τοποθέτηση νομίζω ότι πραγματικά είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Κοινοβουλίου να τοποθετηθεί καθαρά και να αντιταχθεί στη θέση ορισμένων ε, χωρών μελών στο Συμβούλιο, γιατί χρωστάμε, το χρωστάμε αυτό στους εκλογείς μας, οι οποίοι αυτό αναμένουν από μας. Δεύτερο, θεωρώ ότι η μετανάστευση μέσω της Μεσογείου πρέπει να γίνει η εξαίρεση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε άλλα μέσα, άλλα εργαλεία για να μπορεί να γίνεται η μετανάστευση αυτή. Τα συμβάντα αυτά τα οποία ανέφερε και ο εισηγητής είναι ανθρώπινες τραγωδίες μεγάλου μεγέθους και πρέπει να παρακολουθήσουμε και τις ε, επιχειρήσεις της Frontex ε, στον διάδρομο του Γιβραλτάρ και γι' αυτό νομίζω ότι στην έκθεση πρέπει κυρίως να μιλήσουμε για την διάσωση ανθρώπινων ζώων. Αυτό πρέπει να μπει στο προσκήνιο της εκθέσεως. Γι' αυτό ευχαριστώ τον εισηγητή για τις καλά μελετημένες τροπολογίες του, για την σωστή ένταξη στο κείμενό του του δικαιώματος της μη επανεισδοχής, δηλαδή της μη ε, αποστολής στη χώρα προέλευσης και Αυτά τα ε, περιλαμβάνει και στην τροπολογία 1. Θετικό επίσης είναι, αντίθετα με την πρόταση της Κομισιόν, η διαγραφή του αρθρού 7.1.ε. Έχω και ορισμένα σημεία κριτικής γιατί αυτή η υποχρέωση διάσωση στην ανοιχτή θάλασσα δεν ισχύει και για παράκτης περιοχές. Αλλά μπορώ να το συζητήσω, δηλαδή, για, ε, κοντά στις ακτές, στη θάλασσα πάντα, ε, θα το συζητήσω αυτό διμερώς με τον εισηγητή για να αποφύγουμε συμβάντα όπως αυτό στα νυχτά της Λαμπεντούσα. Επίσης η επιχειρησιακή συνεργασία με τρίτες χώρες. Θα πρέπει να αποκλειστεί η συνεργασία με τρίτες χώρες όπου υπάρχουν επιφυλάξει για την στάση τους απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Βρίσκω θετικό ότι θεσπίζεται υποχρέωση της Frontex να υποβάλει έκθεση αναδιαιτία στο Κοινοβούλιο. Νομίζω μάλιστα ότι εδώ μπορούμε να σημειώσουμε και ότι οι ενστάσεις κατά της επανεισδοχής πρέπει να καταγράφονται ώστε και μετά από την πάροδο της διετίας να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι θεωρώ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα οι πρόσφυγες να μπορούν να προβάλλουν και ένσταση κατά της εφαρμογής ή μάλλον κατά της παραβίασης της αρχής της μη επανεισδοχής. να δούμε αν ίσως η ένσταση αυτή πρέπει να έχει και ανασταλτικό αποτέλεσμα. Βρίσκω λοιπόν εν τέλει και πάλι ότι πρόκειται για μια καλή έκθεση που θα μας επιτρέψει να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις πολλές αγωνιώδεις ερωτήσεις των πολιτών στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο εδώ μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Βίξτρομ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Κόλλο, γιατί για κάτι πήγοντος χαρακτήρα κειμένου. Και ακόμη πιο επίκαιρο είναι με το τραγωδία στην Αμπεντούζα, είναι τόσο πρόσφατη και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για όλους ότι οι σημερινές πολιτικές δεν λειτουργούν, δεν αποδίδουν. Και ότι πιο πολλά θα πρέπει να κάνουμε σχετικά με το πρόβλημα. Άρα να κάτσουμε και να δούμε που δεν τα πήγαμε καλά, να μην κατηγορούμε άλλους, να τονίσουμε ότι τρίτες χώρες ε, λέμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οπότε, όπως είναι τώρα τα πράγματα. Μου φαίνεται αποκοτευτικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται από κάποια κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να τον χωνέψω αυτό γιατί το πρόβλημα είναι πως τα κράτη-μέλη που γνωρίζουμε επανειλημμένα ισχυρίζονται ότι συντρέχει το εθνική αρμοδιότητα και αρνούνται την ε, επίλυση του θέματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απέκτησε τα απαραίτητα μέσα ε, στις ε, κοινωτικές της υπηρεσίες για να κάνει κάτι για το πρόβλημα και γι' αυτό και εγώ δεν πιστεύω ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτήσει τα εγγύα μέσα πολιτικής, τότε θα αναλάβει τις ευθύνες της. Και τέτοιε τραγωδίες, σαν αυτά, τα πρόσφατα γεγονότα που έγιναν στην Μεσόγειο, στα Μεντούζα, όλα αυτά είναι θέματα ευρωπαϊκά και θα πρέπει επομένω σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίζονται. Δεν ε, είναι σοβαρό τα κρατημέλη να αλληλοκατηγορούνται ε, και να, να, να, να εκτρέπονται, να καταγγέλουν. Είναι ηρωνικό, είναι κινησμό και τέτοιο, γιατί έχουμε τώρα πάνω από 200 οι οποίοι έχασαν τη ζωή του στην Μεσόγειο. Ήδη χαίρεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπα ότι είναι πάρα πολύ καλή και είπαμε ότι οι τροπολογίε του κ. Κοελιό πρόκειται να θωρακίσουν περισσότερο τον κανονισμό. Οπότε και σήμερα το πρωί με μεγάλη μου χαρά μπορώ να σα πω ότι δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την προσέγγιση Κοέλιο. όντω πρόκειται περί άρτια έκθεση. Και θα πρέπει, όχι εκτό από το ΕΛ και το κύριο Κόλλιο, όλοι να είμαστε υπερήφανοι, μια που σήμερα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα κατόπιν των όσων έγιναν. Θεώρησα επίσης ότι θα πρέπει να καθοριστούν ευθύνες εκάστου καλύτερα, η αρχή της ε, μη επαναπρόθεσης και η αποποινικοποίηση των αλλιέων και άλλων προσώπων. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς θα σώσουμε ε, ανθρώπινες ζωές στη Μεσόγειο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η ηθική μας υποχρέωση. Η ηθική υποχρέωση κάθε ανθρώπου να προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μην τους κατηγορούμε αυτούς τους ανθρώπους μην τους ενοχοποιούμε. Έχω κατεβάσει εγώ κάποιες ε, τροπολογίες στο μικρό σχήμα των Σολοκίων Σκόλια, δηλαδή τονίζουμε ότι η συνεργασία με τις τρίτες θα πρέπει να είναι στα πλαίσια του εξασφαλισμού των ανθρωπινών ε, ε, δικαιωμάτων και επίσης όπως την υπόθεση χάρηση θα πρέπει αυτέ οι αρχέ να γίνονται σεβαστές και ότι προσδοκούμε την περαιτέρω συνεργασία για το ζήτημα. Δεν ξέρω, ήταν θέμα ίσως διατύπωσης και δεν κατάλαβα καλά θα έπρεπε να μας πει περισσότερα το Συμβούλιο για την στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει. Γιατί είναι αυτονόητο ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι ήσασταν αρκετά φιλόδοξοι. Οπότε παρακαλώ περιμένω να ακούσω περισσότερο γιατί είναι πάνω περισσότερο από σημαντικό να κινηθούμε. Δεν είναι δυνατόν να ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια θέση. Να βρούμε κατάλληλα μέσα πολιτική και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά για την καλή δουλειά που κάνατε και που βελτιώνετε κι άλλο το κείμενο της Κομισιόν ώστε έτσι θα μπορέσουμε να δούμε και τις τροπολογίες σας για τα θέματα του χώρου ασφαλείας, ε, την αρχή της μη επαναπροώθησης, τον μηχανισμό της αλληλεγγύης και τη δυνατότητα ε, να μπορέσουμε να στείλουμε και σκάφος για διάσωση στην ανοιχτή θάλασσα. Έχουμε κάποιες ε, αμφιβολίες όμως για το κατά πόσον οι επιχειρήσεις της Frontex στη θάλασσα θα συνάδουν πλήρως με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι υπάρχουν θέματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ε, τα οποία βρίσκονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας ευχαριστώ, αλλά και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η δική σας δεν επιλύουν το βασικό θέμα. Πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά αποτελεσματικά και στην ανοιχτή θάλασσα. Η απόφαση χέρση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει σαφέστατα ότι η αποβίβαση ατόμων σε τρίτες επιτρέπονται βάσει συγκεκριμένων κανόνων διεθνούς δικαίου, που είναι ότι μπορεί να γίνει αποβίβαση μόνο οι συγκεκριμένες συνθήκες του καθενός αξιολογηθούν χωρίς κανένα περιορισμό, μπορεί να γίνει μόνο εάν ενημερωθούν πλήρως ε, τα άτομα για τη διαδικασία, αν έχουν πρόσβαση σε διερμηνέα και εάν υπάρχει πρόσβαση σε νομική συνδρομή. Αλλά πέραν της ενημέρωσης για το χώρο της αποβίβασης, Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνονται πλέον στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο σχέδιο έκθεσης. Και αν δεν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, τότε σίγουρα δεν υπάρχει σύμπνοια με την απόφαση του δικαστηρίου. Και φυσικά ε, ελοχεύει ο κίνδυνο να παραβιάσουμε και το διεθνέ και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εμεί ω πράσινοι έχουμε πει ότι εν γέννη έχουμε αμφιβολίε για το κατά πόσον είναι δυνατόν να παρέχουμε τέτοιε εγγυήσει επί ενό σκάφου στην ανοιχτή θάλασσα. Αλλά εάν η πλειοψηφία του του Κοινοβουλίου θεωρεί ότι θα πρέπει ε, να υπάρχουν και να ευνοούνται αυτές οι επιστροφές, τότε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι γίνεται σεβαστή τουλάχιστον η απόφαση του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι δεν υπάρχει παραβίαση διεθνούς δικαίου για την έρευνα και τη διάσωση συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή και οποιονδήποτε άλλον είπε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά αυτά τα μέτρα, ιδίως μετά τη Λαμπεντούζα και επειδή έχουμε βιώσει και αντίστοιχες καταστροφές, όχι ίσως τόσο μεγάλης κλίμακας και σε άλλες χώρες, θα πρέπει ε, να ε, προσπαθήσουμε να το επιβάλλουμε εμείς διότι φαίνεται ότι κάποιες χώρες θα προσπαθήσουν να σταματήσουν αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστές οι χώρες, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Μάλτα. Και είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, είναι απαράδεκτο να ε, φτάνουν σε τέλμα αυτές οι καταστάσεις ε, στο Συμβούλιο μετά από αυτή την καταστροφή. Όλοι λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Η Ιταλία έκανε έκκληση για περισσότερη ευρωπαϊκή υποστήριξη. Πώς μπορούν λοιπόν, πώς μπορεί το Συμβούλιο να μπλοκάρει μια, ένα τόσο σημαντικό θέμα της έρευνας και της διάσωσης και τους σχετικούς κανόνες. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις της Frontex είναι στην πραγματικότητα επιχειρήσεις έρευνα και διάσωσης, θα ήθελα να επαναλάβω το ερώτημα το οποίο έχω θέσει και επανειλημμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσες από τις ε, επιχειρήσεις ε, επιτήρησης συνόρων τελικώς καταλήγουν να είναι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία είτε ποσοστά είτε αριθμητικά συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε και κάποιες αμφιβολίες για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποβίβαση σε τρίτες χώρες ως ε, την προτιμόνεμη λύση, διότι αυτή η αποβίβαση θα πρέπει να γίνεται πάντα στον πλησιέστερο ασφαλές σημείο και θα πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια από την, ε, με βάση την αρχή της μη επαναπροώθησης. Και δεν θα πρέπει να θεωρείται διάσωση όταν κάποιος τους ε, ε, φτάνει σε ένα λιμάνι τρίτης χώρας. Πρέπει να φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί στο ασφαλέστερο σημείο. Και αν είναι αυτό κράτο μέλο, τότε θα πρέπει να πάει σε αυτό. Όσον αφορά το μηχανισμό τη αλληλεγγύη, σαφώ υποστηρίζουμε το μηχανισμό αλληλεγγύη που προτείνει ο, ο Είναι ένα πρώτο βήμα για να υπάρχει περισσότερο καταμερισμό ευθυνών μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ήθελα να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προ αυτή την κατάσταση. Τα κράτη-μέλη στη νότια πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται σίγουρα περισσότερη υποστήριξη και επομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει να τους βοηθήσουμε για να διασώζουν πρόσφυγες, ε, θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα επαναγκατάστασης και θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα για να εφαρμόζεται διαφορετικά κανόνες του Διβλίνου 2 ε, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να βοηθηθούν, υπάρχουν πάρα πολλές ε, παραβιάσεις και στην Ιταλία και στην Ελλάδα κατά ετούν τον άσυλο και θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ερωτήσεις μου. Κυρία Βερυζιά. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Τα ουσιαστικά τα είπαμε άλλωστε. Ε, αντικαθιστώ λίγο τη συνάδελφο την Κορνέλια Ένση, η οποία είναι ισχυώδη συζητήτρια για το θέμα αυτό. Και ομολογώ, κύριε Σιγητά, ότι δεν έχω διαβάσει ακριβώ τι θέσει σα, επομένω είμαι λίγο σε δύσκολη θέση. Ωστόσο, από αυτά που άκουσα και κυρίως από τον προσανατολισμό της ε, πρότασής σας, αυτά που κατάλαβα λοιπόν, με βρίσκουν σύμφωνοι διότι θεωρώ ότι στον τομέα αυτό είμαστε μπλεγμένοι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, όλοι μαζί για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο. Η στάση κάποιων κρατών μελών που είναι αυτά τα οποία ε, συνήθως ε, κάνουν περισσότερο έκκληση για την ευθύνη και την αλληλεγγύη και προσπαθούν να μας επιβάλλουν την άποψή τους για τους πιο ευάλωτους και τα ε, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες. Υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ αυτών που κάνουν και, αυτά που, και αυτών που λένε. η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματι... αποδεδειγμένα δεν έχει κάνει τίποτα και ξέρουμε ότι μας ενδιαφέρει κυρίως η ευθύνη των κρατών μελών ε, και υπάρχει και ευθύνη φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά με βρίσκουν σύμφωνοι. Θα ήθελα να επιμείνω σε κάποια σημεία τα οποία αναφέρθηκαν μεν, αλλά τα θεωρώ σημαντικά δε. Συνεργασία με τρίτες χώρες, η οποία θα πρέπει να αποκλείεται όπως είπατε και εσείς, όταν τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Υπάρχουν κάποιες χώρες με τις οποίες υπάρχουν συμφωνίες επανεισδοχής ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διμερές επίπεδο. Η συνάδελφος Σίσκα Κέλλερ επέμενε για κάποια σημεία τα οποία τα έχει θίξει και ο εισηγητής του ΟΗΕ για το θέμα αυτό την ανάγκη να υπάρχουν πληροφορίες ε, ε, για την ε, χώρα της αποβίβασης, η ανάγκη ύπαρξης διερμηνίας, νομικής συνδρομής. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία είναι ουσιαστικά και θεωρώ ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί ώστε να υπάρχει έστω μια κάποια ελάχιστη συνέπεια για το θέμα αυτό, διότι όπως είπατε και εσείς κύριε Σιγητά, πρόκειται για ανθρώπινες ζωές η Λαμπεντούσα θα πρέπει να μας χρησιμεύσει ως αποκάλυψη, διότι είναι το πιο σημαντικό δυστύχημα των τελευταίων ετών. Ένα δράμα το οποίο έλαβε χώρα στα 600 μέτρα από την ακτή. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δίστασαν να τρέξουν σε βοήθεια ανθρώπων ε, ε, των οποίων κινδύνευε η ζωή με βάση την Ιταλική νομοθεσία και όλα αυτά φυσικά είναι απαράδεκτα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βελτιώσουμε τα θέματα και να μπορέσουμε να αναστρέψουμε και τη θέση του Συμβουλίου. Ο κύριος ε, Κίρκοπ. Καταρχά, ζητώ συγγνώμη. Το Κοινοβούλιο, όπω ξέρετε, έχει πάρα πολλά να κάνει τη σημερινή μέρα. Αλλά θέλω να σα πω παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην καταλήξουμε σε μια στάση υποκριτική η πολιτική μας ομάδα είναι ανοφαντών υπέρ τέτοιων πρωτοβουλειών. Αλλά το πρόβλημα μας είναι το εξή. Πρώτα πρώτα μας κατηγορούν κάποιες χώρες ότι δεν κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά. Όμως το Συμβούλιο συνεδρίαση, κατόπιν συνεδρίασης υπάρχουν κάποιες προτάσεις από την Frontex για δραστηριότητες στη Μεσόγειο κλπ. Στο Συμβούλιο λοιπόν τα κράτη-μέλη, ιδίως τα κράτη εκείνα που βρέχονται πριν Μεσόγειο, προτάσουν ενστάσεις. Ισχύει ότι υπάρχουν προβλήματα και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Και είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι και οι άλλοι εδώ βουλευτές και εκπρόσωποι των Ευρωπαίων αισθανόμαστε αμηχανία. Προβληματιζόμαστε από αυτά όλα τα γεγονότα τα οποία γίνονται στις ακτές μας, στις θάλασσές μας. Είναι αποτρόπια αυτά τα οποία έγιναν με αυτά τα σκάφη και με τους θανάτους προήψαν. Πρόκειται για στίγμα το οποίο θα πρέπει να το βοηθούμε και να το διαχειριστούμε κατεπηγόντως και προσεκτικά. Επομένως, νομίζω ότι τα κρατημένη θα πρέπει να συζητήσουν για να αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν και πώς να σώσουν αυτές τις ε, ζωές. Όμως πάλι θα πρέπει να έχει πιο δυναμική πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις πηγές αυτών των προβλημάτων. Γιατί μιλούμε για συνεργασία με τρίτες χώρες για να αποτρέψουμε τους μετανάστες να μην ε, κάνουν αυτές τις, ε, αυτά τα, τα, τα, τα επικίνδυνα ταξίδια. Θυμάμαι από μία ή δύο θητείες είχαμε πάρα πολύ προβληματιστεί με την Λιβύη γιατί τη διάφορα δικτατορικά καθεστώτα, φόρτωναν σχεδίες και τις στέλναν προς τη Λαμπεδούσα και την ε, Μάλτα. Ήταν εντροπή. Και δεν ίσχυσε καμία ιδιαίτερη πίεση σε αυτά τα καθεστώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μόχλους πίεσης. Έχουμε συμφωνίες ε, σύνδεσης, χρωματοδοτικές ε, άλλε συμφωνίε οικονομική υποστήριξη. Α τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Α αναβαθμίσουμε τη δράση μα κατά του οργανωμένου εγκλήματο. Γιατί αυτέ οι μαφίε εκμεταλλεύονται του μετανάστε και δίνουν δεκάρα για το πού θα ζήσουν ή αν θα πεθάνουν. Και του ζητάνε τρομερά ποσά για να τους βοηθήσουν. Πάρα πολύ κακά όλο. αυτό. Άρα θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερο. Και θέλουμε έναν πιο συνεκτικό, έναν πιο ουσιαστικό διάλογο για τα θέματα της μετανάστευσης, της κινητικότητας και της ασφάλειας για τα σύνορά μας, για τη διαχείριση αυτών. Έχω βαρεθεί να ακούω συγγνώμες, θλίψη, αλλά καμία πρόταση. Πρέπει επομένω να δώσουμε στην προτεραιότητα σε αυτό το πρόβλημα. Και όποτε υπάρχει εμπλοκή από Συμβούλιο και κρατημέλη, τότε και εμεί θα πρέπει να κατονομάζουμε ακριβώ ποια είναι τα... ποιοι είναι αυτοί που δεν αφήνουν να λυθούν το πρόβλημα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συνάδελφοι με κάλυψαν. Και εγώ συμφωνώ με όλα όσα άκουσα. Να προσθέσω μόνο το ότι ευχαριστώ τον Κάρλος. Είναι εξαίρετη η έκθεσή του. Είμαι βέβαιος επειδή τον έχω μάθει για τα καλά ότι θα τα καταφέρει. Θα μπορέσει να πείσει όλες τις πολιτικές ομάδες και ότι το αποτέλεσμα θα είναι μια εξαιρετική έκθεση που θα καλύψει τους πάντες. Ε, ε, ε, η κυρία Γκόμες. Πολύ σημαντικά όλα αυτά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ με όλα σου άκουσα. Επίσης, σύμφωνα με αυτούς που είπαν ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πρωτοπόρο σε αυτόν τον αγώνα. Δεν πρόκειται για πρόβλημα μετανάστευσης. ή το πρόβλημα αυτών που είναι πρόσφυγες και που ζητούν άσυλο. Κάποτε μιλούσαμε για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρώπη, για τις μεταναστευτικές ροές κλπ. κλπ. Όμως μετά ήρθε η κρίση. Η κρίση έγινε γνωστή και στις χώρες των μεταναστών. Και είδατε ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που προσπάθησαν στην Ευρώπη και πνιγήκαν στη Λαμπεντούσα και στην ε, Μάλτα. Επρόκειτο για πρόσφυγες από τον πόλεμο της Συρίας, από την σύραξη την εμφύλια στην Σομαλία. Πρόκειται για άτομα τα οποία προσπάθησαν να γλιτώσουν την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους σε Ερυθρία και Σουδάν. Να επομένως, Καταμίζω ένα λόγο γιατί στα πλαίσια αυτής της οδηγίας να είμαστε εμείς πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή, να απαιτήσουμε χώρες όπως η, Ιταλία που ποινικοποιεί αγίνους προς να σώσουν αυτούς που πνίγονται στη θάλασσα να καταργήσουν αυτές τις ποινικέ διατάξεις που αντιβαίνουν στα ανθρωπινά δικαιώματα. Αντιστρόφως, θα έπρεπε στην οδηγία να ποινικοποιήσουμε τη συμπεριφορά εκείνων που εκουσίως που αρνούνται να βοηθήσουν αυτούς που διατρέχουν τον κίνδυνο ζωής. Ακόμα και δεν είναι υπάλληλοι της Frontex, ακόμα και είναι υπάλληλοι εθνικών διοικητικών αρχών. Επίσης, κάτι για τον κύριο Κέρκοπ. Μας είπε για το τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με της χώρες προέλευσης και είπε ότι δεν είναι αυτή η οικονομική μετανάστες. Είναι πρόσφυγες, ζητάνε άσυλο αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, να μιλάμε σήμερα για τη Λιβύη, είναι παράλογο. Θυμάστε τι έκανε η Λιβύη του Καντάφη. Εξεβίαζε την Ευρώπη με τους μετάστες που έστειλαν στην Ευρώπη. Όντως θα πρέπει να δούμε και τις άλλες πολιτικές, οι οποίες όμως αποδίδουν. Όμως, προσοχή να μην έχουμε στρεβλωτικά αποτελέσματα, όπως με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είδατε τι γίνεται στην Ερυθρέα και στην Αιθιοπία. Ο κόσμος από εκεί προσπαθεί να ξεφύγει. Και εμείς τι κάνουμε. Α, και στη Σομαλία, σε κάτι υποδιάλυση. Στην Αιθιοπία. Δεν έχουμε σωστή θέση. Και για τη Λιβύη, να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ είμαι η μόνιμη εισηγήτρια για τη Λιβύη. Το είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Από εκεί έφυγε το σκάφος αυτό που μετά βρίσκεται στη Λαμπεντούζα. Από μία πόλη στη Λιβύη που είναι από τις πιο ασφαλείς που έχει μια τοπική φυλακή που λειτουργεί άψογα. 50 χιλιόμετρα μακριά από αυτή τη Λιβυκή πόλη όμως έχουμε ε, μια ανεξέλεγκτη ζώνη, no man's land. Επομένω η αποστολή τη Ευρώπη ε, εν προκειμένου είναι κάτι να κάνει σε σχέση με την, ε, την ΚΕΠΑ. Θα πρέπει να βρεθεί μια δομή ασφάλειας. Δεν υπάρχει βέβαια στη Λιβύη. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση Και δεν λέω μόνο τη χώρα του κύριου Κέρχοπ, αλλά και η Ιταλία και η Γαλλία τι κάνουν. Αντιτίθενται στο να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες δομές ασφαλείας ή στην Λιβύη. Δεν έχουν αυτά που χρειάζεται, δεν έχουν στρατό. Δεν, δεν είχε τέτοια πράγματα η Λιβύη, κάτι προεδρική φρουρά, πρετοριανούς είχε μόνο. Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, Υπουργείο Εσωτερικών, εκεί θα πρέπει να βοηθήσουμε να αποκτήσουμε το υλικό. Το υλικό το αποκτούν, αλλά δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Γιατί δεν έχουν ούτε στρατό ούτε αστυνομία. Οπότε Έχουμε τις πολιτιοφυλακές που δρούν εκεί. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς, να έχουμε ολοκληρωμένες πολιτικές, σφαιρικές. Είδατε τώρα ποιες είναι οι συνέπειες της αποτυχίας μας σε άλλες πολιτικές. Επομένως, μπράβο, θα υποστηρίξω τη δουλειά του Κάρλος Κόλλιου αλλά να αναβαθμίσουμε την έξαρση του και να ζητήσουμε την ποινικοποίηση εκείνων οποία αρνούνται να σώσουν τα πρόσωπα αυτά που διατρέχουν κίνδυνο. και προκύπτει ότι σε κάποια κρατημέλη, όπως και στο δικό μου που είναι η πατρίδα του Κάρλος Κόλλιο, θέλουν με καινούργια νομοθεσία να ακυρώσουν κάποιες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το άσυλο και την προστασία των προσφύγων. Ετέθησαν κάποιες ερωτήσεις. Ήρθε η ώρα το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Απαντή να απαντήσουν. Θέλετε να απαντήσετε. Όχι. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Δεν μία αντίδραση. Ωραία. Να δώσουμε τον λόγο στον εισηγητή. Κύριε Κόγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω του συναδέλφους ε, για την ευρεία υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Να πω στη Φρανσίσκα Κέλλερ ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει, μεν, αλλά μπορεί να καταλάβει ίσως ότι όταν ε, απαγορεύουμε την επιστροφή στην ανοιχτή θάλασσα, επιλύουμε τμήμα του προβλήματος, όχι όλα τα προβλήματα, αλλά τμήμα του προβλήματος και δεν έχουμε νομικό περιθώριο να ε, τους πάμε αλλού, κυρίως σε χωρικά υδατά άλλης χώρας. Να σας διαβεβαιώσω ότι οι επιχειρήσεις της Frontex θα ε, λειτουργούν με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό το στόχο έχει η εκθεσή μου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από την Προεδρία να διαβιβάσει ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο. Το μήνυμα είναι σαφές. Μην είστε υποκριτές. Εάν τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο πραγματικά ανησυχούν για τις ανθρώπινες ζωές, Τώρα είναι η ευκαιρία να αποδείξουν ότι μιλάνε σοβαρά. Και κατά την άποψή μου, εάν το Συμβούλιο θέλει πράγματι να σώσει ανθρώπινες ζωές, έχει αυτή την ευκαιρία στη διάρκεια αυτή τη Προεδρία να καταλήξει σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εγκρίνει τη συγκεκριμένη νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν. Αυτό σημαίνει πριν από το Δεκέμβριο του Τρέχοντο. Εάν το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να το κάνει αυτό, όπω. Ε, αντιλαμβάνομαι από αυτές τις φρικτές δηλώσεις που διαβάσαμε στον τύπο αυτή την εβδομάδα, μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι ψεύδονται όταν παριστάνουν τους λυπημένους και τους ανήσυχους για τις τραγωδίες που βλέπουμε καθημερινά στη Μεσόγειο. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να αποδείξουν ότι μιλούν σοβαρά. Σας παρακαλώ λοιπόν συμφωνήστε μαζί μας πριν το Δεκέμβριο του 2013. Απόλυτα κατανοητό, σαφέστατο το μήνυμά σας. Να περάσουμε λοιπόν στην προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών 19 Οκτωβρίου, εξέταση τροπολογιών εδώ στην Επιτροπή Λίμπε στις 14 Νοεμβρίου. Ωραία. Επιτρέψτε μου τώρα να διακόψουμε για 10 λεπτά, διότι έχουμε συνεδρίαση συντονιστών προγραμματισμένη για τις 12. Να μπορέσουν να έρθουν λοιπόν και οι υπόλοιποι συντονιστές. Δέκα λεπτά ένα διαλυματάκι και ε, θα συνεδριάσει οι συντονιστές και κλεισμένων των θυρών στις 12.